Let's start, ladies and gentlemen. Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι αν θέλετε. Κάποιες πληροφορίες για καταρχήν. Έχουμε τις εξής, μάλλον έχουμε τις εξής γλώσσες που δεν μεταφράζονται, δανικά, σουηδικά, φιλανδικά, λα, λετονικά, σλοβενικά, σλοβακικά, βουλγάρικα, εστονικά, τσέχικα. Έχουμε τις γλώσσες μονάχα των πλήρων μελών της Επιτροπής και η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη σε διάταξη. Αν υπάρξουν μέχρι στο τέλος παρατηρήσεις, ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 13 Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτεμβρίου και 25-26 Οκτωβρίου 2010. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις στο τέλος της συνεδρίας θα κάνω τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις. Σημείο 4 της τη διάταξης. Μέθοδη πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης βάσει του συστήματος Galileo. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στη λεγόμενη Public Regulated Service, την ε, δημόσια κυβερνητικού χαρακτήρα υπηρεσία, μεταξύ των πέντε υπηρεσιών που θα προσφέρει τον Γαλιλαίο. Μία από αυτές είναι η Public Regulated Service, η λεγόμενη κυβερνητική υπηρεσία η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από φορεί οι οποίοι έχουν τύχει διαπίστευτη από τι αντίστοιχε κυβερνήσει, αφορά επικοινωνίε ευαίσθητου χαρακτήρα και απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συνέχεια παροχή υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή, η λεγόμενη PRS, είναι μια υπηρεσία που έχει εφαρμογέ οι οποίε είναι ευαίσθητε από πολιτική και στρατηγική έποψη. Για του λόγου αυτού, για λόγου ασφάλεια, και εμπιστευτικότητα θα πρέπει να την χάνει αυστηρής επιτήρησης και ελέγχου. Λόγω των χαρακτηριστικών λοιπόν αυτής της υπηρεσίας PRS χρειάζεται επακριβής καθορισμός των κανόνων πρόσβασης σε αυτή την υπηρεσία μέσω ενός νομοθετικού κειμένου. Το κείμενο το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα το οποίο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις ε, αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ικανοποιεί αυτά τα προαπαιτούμενα. Η πρόταση της Κομισιόν εστιάζεται σε τρία κύρια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα. Περιλαμβάνει μια σειρά από γενικές αρχές σε σχέση με τους κανόνες πρόσβασης στην υπηρεσία PRS. Δεύτερον, περιλαμβάνει την υποχρέωση για τα κράτη-μέλη, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία PRS, να καθορίσουν μια αρμόδια αρχή για την υπηρεσία PRS, η οποία παρακολουθεί την κατασκευή, την ε, αποθήκευση και τη χρήση δεκτών PRS, βέβαια τηρώντας ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές. Και τρίτον, η εισαγωγή στο νομοθετικό κείμενο προϋποθέσεων για την κατασκευή και την εμπιστευτικοποίηση των συσκευών PRS. Η πρόταση προβλέπει κεντρική διαχείριση ορισμένων στοιχείων σε κοινοτικό δηλαδή επίπεδο, διότι αυτό είναι και εφικτό και επιθυμητό. Σε ό,τι αφορά τώρα άλλα στοιχεία της πρότασης, φαίνεται πιο πρόσφορο να ακολουθήσουμε μια αποκεντρωμένη μορφή διαχείρισης στα κράτη-μέλη, τα οποία είναι στην καλύτερη θέση για να φέρουν σε πέρας αυτό το καθήκον, παρά το γεγονός ότι η υποδομή παραμένει στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι η πρόταση αυτή είναι το πόρισμα εντατικής προπαρασκευαστικής εργασίας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια τεχνικού χαρακτήρα πρόταση και όχι πολιτικού χαρακτήρα πρόταση. Δεν είναι ο στόχος μας να ρυθμίσουμε τις δυνητικές εφαρμογές της υπηρεσίας PRS, αυτές καθεαυτής, αλλά μονάχα τους κανόνες πρόσβασης στην υπηρεσία PRS. Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Συμβουλίου ήταν ιδιαίτερα θετική και ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει αυτό το νομοθέτημα και θα το διεκπαιρεώσει ταχαίως και θα είναι σε θέση να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό την πρόταση της Κομισιόν. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια απόφαση την άνοιξη του 2011. Διότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και μια βάση για να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις σε επίπεδο βιομηχανικό για την κατασκευή των δεκτών οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους δέκτες. No. Okay. Uh, thing. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Άκουσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις συχνότητες του Γαλιλαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει κάποιες συχνότητες, από ό,τι φαίνεται όμως χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι δορυφόροι τις συχνότητες αυτές. Είναι σοβαρό από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσετε εσείς άλλες συχνότητες, τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά, πώς θα την ξεπεράσουμε. και σε ποιο βαθμό η δράση και και, και η, εξωτε, η υπηρεσία εξωτερική δράση θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό μέσω του Γαλιλαίου. Ευχαριστώ κυρία Τσέκ. Δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη ερώτηση. Καλώς. Ο εκπρόσωπος Επιτροπής έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για την Κίνα. Ξέρετε ότι από το 2004 υπάρχει μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες μας χαροποιεί η συμφωνία αυτή γιατί καθορίζει και ρυθμίζει σωστά το τι θέλει κάθε πλευρά. Με την Κίνα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε μια συμφωνία μεν από το 2003, αλλά εξακολουθούν οι συζητήσεις γύρω από το θέμα των συχνοτήτων. Είναι σοβαρό το θέμα ο κύριος Μπαρόσο έγραψε μια επιστολή στον ομόλογό του, τον Πρωθυπουργό της Κίνας. Και η απάντηση που δόθηκε είναι ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα σε τεχνικό επίπεδο. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν έχουμε ε, προχωρήσει. Ανησυχούμε γιατί το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί σύντομα και θα ήθελα και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας βοηθήσει να ρυθμιστεί εν πάση το θέμα αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Είναι κάτι το οποίο αφορά και τις λεγόμενες public regulated services αλλά και γενικότερα το ευρύ Επαναλαμβάνω ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα και αναζητούμε μία λύση. Η δεύτερη ερώτηση believes that each member state will decide independently how to use the PRS uh, in this uh, area of competence. But we think also Λοιπόν, το θέμα της, του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί. Η συνεργασία α, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και της Δράσης ΚΕΠΑ είναι μια συνεργασία την οποία επιθυμούμε σφόδρα και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του συστήματος αυτού με τρόπο που να είναι θετικός εν πάση περιπτώσει. Thank you very much. Mr. vielen Dank. Mir Σας ευχαριστώ. Μου ήρθε τώρα μια ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμά σας. Πότε νομίζετε ότι το, το πρόγραμμα, μάλλον πότε θα έχουμε προχωρήσει αρκετά ώστε να τεθεί το πρόβλημα στην πράξη. Πόσα μέρη ε, θεωρείτε ότι θα είναι ενδιαφερόμενα. Έχουν ήδη δηλώσει όλοι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσει για τη χρήση του μέσου κλπ. Thank you. We have made... Προχωρήσαμε σε μια ανάλυση εδώ και λίγο καιρό, η οποία όμως δεν είναι πλέον ενημερωμένη. Τα κράτη-μέλη πάντως ζήτησαν υψηλά επίπεδα συνεργασίας. Προς το παρόν περιοριζόμαστε σε ομάδες εργασίας σε κάθε χώρα ή και σε περιφερειακό επίπεδο για να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται. Υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον. Προετοιμαζόμεθα επίσης και προλιένουμε το έδαφο σε τεχνικό επίπεδο για να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει σωστά και ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία προκήρυξης ε, για την κατασκευή των ε, νέων δεκτών. Ελπίζουμε να επιταχύνουμε τα πράγματα έτσι ώστε να καταστεί λειτουργική η παροχή αυτής της υπηρεσίας από το 14 και μετά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λούιζινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω κάποιος άλλος να μην έχει θέσει ήδη την ερώτησή μου και αν ναι, αγνοήστε την, αλλά είναι η εξής. Τονίζεται ξανά και ξανά ότι το Γαλιλαίο είναι μη στρατιωτικό πρόγραμμα υπό μη στρατιωτικό πολιτικό έλεγχο δηλαδή. Τώρα, στο 2010-550 της Κομισιόν, βλέπω μια ε, γραφική παράσταση που δείχνει 50% στρατιωτική χρήση του συστήματος. Πώς συμβαδίζουν αυτά με τις αρχικές δηλώσεις που γέννηκαν για το θέμα. Και εδώ έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Βλέπω σε ένα περιοδικό Technology Review που επικαλείται τον Γερμανό Διευθυντή ε, Αεροδιαστημικής Έρευνας να λέει ότι η συμμετοχή της Κίνας στο Γαλιλαίο λόγω της στρατιωτικής, ε, ε, αποτράπηκε λόγω της μελλοντικής στρατιωτικής χρήσης του ε, συστήματος ενώ με τη συμμετοχή αυτή θα ήταν πολύ σημαντικό, σημαντική μείωση του κόστους για την Ευρώπη. Πώς συμβαδίζει αυτό με το γεγονός ότι χρηματοδοτείται η κατασκευή του συστήματος από μη στρατιωτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτη ερώτηση. Τον Οκτώβριο στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύθηκε έκθεση επικαλούμενη πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δήλωνε ότι θα κοστίσει ακριβότερο το σύστημα μεταξύ 1,5 και 17 δισεκατομμύριων ευρώ. Και ακόμα χειρότερα, λέει ότι ο Γαλιλαίος ποτέ δεν πρόκειται να είναι κερδοφόρος και ότι κάθε χρόνο θα προκαλεί ζημία 750 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Μήπως είναι καλύτερο να το θάψετε το σύστημα. Thank you, Uh... Ευχαριστώ πολύ. Κύριο σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα σας υπενθυμίσω ότι βάσει του κανονισμού 683 του 2008 αναφέρεται στην ε, δεύτερη αιτιολογική αναφορά ότι ο στόχος του Γαλιλαίου είναι να δημιουργήσει την ε, πρώτη υποδομή για ραδιοπλοήγηση και εντοπισμό ε, για πολιτικούς σκοπούς καταρχήν. Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος Γαλιλαίου. Αυτό τονίστηκε επίσης από το Συμβούλιο σε πολλές ευκαιρίες. Μόλον τούτο, το γεγονός ότι η αποστολή του Γαλιλαίου είναι κυρίως μη στρατιωτική, πολιτικού χαρακτήρα δηλαδή, αυτό δεν αποκλείει την δυνητική χρήση για στρατιωτικούς σκοπούς. Παρά το γεγονό ότι το Γαλιλαίο είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα πρόγραμμα, σε τεχνικό επίπεδο οι υπηρεσίε που παρέχονται από τον Γαλιλαίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αποστολέ οι οποίε έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των κρατών μελών. Σε πολιτικό επίπεδο, <clears throat> πιστεύουμε ότι αναπρόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει ποια θα πρέπει να είναι η χρήση την οποία θα κάνει του συστήματος αυτού, του συστήματος Γαλιλαίου. Ως εκ τούτου, σε σχέση με το θέμα της ε, μη στρατιωτικής ή στρατιωτικής χρήσης, <clears throat> το θέμα ήταν αυτό το οποίο σας ανέφερα για το κόστος και τον προϋπολογισμό που είναι το τρίτο ερώτημα που θέσατε. Θα ήθελα να παραπέμψω την, την αξιότιμη κυρία Βουλευτή στο επικείμενο έγγραφο το οποίο θα δημοσιεύσει η Κομισιόν, την ενδιάμεση αναθεώρηση λοιπόν για το θέμα αυτό. Υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στα κρατημέλη, ιδίω στη Γερμανία το φθινόπωρο, επί τη βάση μια έκθεση από το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνα. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτή την έκθεση. Απλώ σα παραπέμπω στην επικείμενη ανακοίνωση τη Κομισιόν σε σχέση με την ενδιάμεση ε, αναθεώρηση του προγράμματος Γαλιλαίου. Φυσικά, έχουμε ενώπιον μας ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών που αποτελεί τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Ήταν ένα από τα σχέδια προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων. και τα αριθμητικά αυτά ποσά των 700 εκατομμύριων το χρόνο που αναφέρθηκαν αφορούν την συντήρηση του συστήματος. Δεν συνάπτονται με τα έσοδα ή τα τέλη τα οποία μπορούν να συλλεγούν από το σύστημα αυτό. Απλώς αναφερόμαστε στην υποδομή, στην συντήρηση της υποδομής για το σύστημα Γαλιλαίος. Το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, <clears throat> θυμίστε μου, μιλούσατε για την Κίνα. Νομίζω ότι εν μέρει απήντησα για το θέμα της Κίνας. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις συχνότητες που χρησιμοποιεί η υπηρεσία PRS, διότι οι Κινέζοι χρησιμοποιούν και αυτοί το ίδιο κομμάτι του ραδιοφάσματος. Εμείς ήδη από το 2003 προσπαθήσαμε να επιλύσουμε με μια συμφωνία το θέμα αυτό αλλά αυτή η συμφωνία έχει γίνει με διαφορετικές, με ένα, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, με διαφορετικές υποθέσεις από ό,τι ε, συμβαίνει τώρα. Γιατί τότε ο Γαλιλαίος ήταν μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Και εκεί ήταν καλόδεκτη η συμμετοχή και η συνεργασία της Κίνας. Αλλά το 2008 η Κομισιόν με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησε στο ότι το σχέδιο Γαλιλαίος δεν θα πρέπει να τύχει χρηματοδότηση από καμία τρίτη χώρα, όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα, πρέπει να χρηματοδοθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σενάριο λοιπόν του 2003 δεν είναι πλέον έγκυρο και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία ε, ελέγχθησαν ότι η Κίνα θα ήθελε ίσως ή θα μπορούσε κτλ. Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφώς. Αποκλειστικός κύριος του σχεδίου είναι η θα μπορουσε τα λοιπά. τωρα τα πραγματα ειναι παρα πολυ Ένωση και η Κομισιόν το διαχειρίζεται εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much for for Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν βλέπω άλλους εδώ ευρωβουλευτές να θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Καλώς λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως σήμερα. Στρατηγικά μέσα αερομεταφορών, ένα μέσο για διαχείριση των κρίσεων και ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες εδώ με τις παρουσιάσεις τους και θα πάρουν μέρος και στη συζήτηση. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον πλήρχο Ιωάννη Παυλόπουλο, διοικητή του Κέντρου Στρατηγικών Μέσων, τον κύριο Ρούσο, τον Μπρούνο Καντέα, του Τμήματος Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, τον ταξίαρχο Βιτσέντζο Πούρη, του στρατιωτικού επιτελείου και τον κύριο Δημήτριο Μουτσιάκη, υπεύθυνο προγράμματος Ευρωπαϊκού Στόλου Αερομεταφορών και περιμένουμε να έρθει ακόμα ο Πέτερ Μπίλινγκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, προτείνω να γίνουν δύο τράπεζες συζητήσεων ουσιαστικά. Δύο-τρεις ομιλητές θα αποτελούν το πρώτο και άλλοι δύο-τρεις το δεύτερο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Άστον, η ύπατη εκπρόσωπος για εξωτερικές υποθέσεις, διόρισε στις 2 Δεκεμβρίου τον Αγκοστίνο Μιότσο υπεύθυνο για τη διαχείριση κρίσεων στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε τον κύριο Μιότσο σε μία από τις επόμενες συναντήσεις της υποεπιτροπής μας. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τους τρεις ομιλητές, τους τρεις πρώτους, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Ρουτσέαο και τον κύριο Κατά, 10 λεπτά το πολύ η παρουσίασή τους έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος παρακαλώ ερωτήσεων από τα παριστάμενα μέλη του Κοινοβουλίου. Κύριε Παυλόπουλε έχετε το λόγο. Mr. Chairman, respectable ladies and gentlemen, my name... Κύριε Πρόεδρε, έντιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέγομαι Ιωάννης Παυλόπουλος από το Ελληνικό Ναυτικό και είμαι στο κέντρο συντονισμού για τις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και στα επόμενα 10-15 λεπτά θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση σε σχέση με τον ΦΟΡΕ, το Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών και τη λειτουργία και τις δραστηριότητε του. το MSCC, δηλαδή το Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσιών Μεταφορών, δημιουργήθηκε το 2004, ανεξάρτητος οργανισμός, με απόφαση του, Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, Εθνικής Άμυνας, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στρατηγικών μεταφορών σε ενέργειες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος και υποστηρίζεται από το, ε, Ευρωπα... από το ελληνικό ε, επιμελητήριο ναυτιλίας. Βλέπετε το οργανόγραμμα τώρα σε αυτή τη διαφάνεια του κέντρου αυτού ως πολυεθνικής εταιρεία. Ο επικεφαλής είναι πλήρχος του ναυτικού, ο οποίος καθορίζεται από την Ελλάδα. Η Ιταλία έχει τον αναπληρωτή διοικητή, αλλά η θέση αυτή παραμένει ακόμα κενή, γιατί συνεχίζεται η διαδικασία κύρωσης των τεχνικών ρυθμίσεων υπό τον αναπληρωτή διοικητή είναι το τμήμα σχεδίου και συντονισμού και το τμήμα παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Οι θέσεις αυτές είναι ανοιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο συντονιστικό κέντρο. Η φυσιολογική θητεία σε αυτά τα κέντρα είναι 2 με 3 χρόνια, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες εθνικές ε, διαδικασίες. Το προσωπικό που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της σελίδος είναι προσωπικό που καθορίζεται από την Ελλάδα. Με συνεργασία και με την Ελληνική Υπηρεσία Ναυτιλίας, την Ελληνική Υπηρεσία Εφοπλιστών, την Γενική Διοίκηση για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και τον ε, Σύμβουλο της, ε, του AMSCC και τον ε, Σύμβουλο από το Λιμενικό Σώμα. Το κέντρο μας παίζει σημαντικό ρόλο σαν λειτουργικό, σαν επιχειρησιακό εργαλείο για να εξασφαλίσει την επιχείρηση, τη διατήρηση και επαναανάπτυξη δυνάμεων. Ο στόχο δεν είναι μονάχα να έχουμε μια γενική εικόνα τη αγορά, αλλά επίση να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε ε, στοιχεία, ε, σε εξοπλισμό για ε, θαλάσσιες μεταφορές και για να μπορούμε να κινητοποιούμε τα κατάλληλα αυτά στοιχεία μέσα, αυτά σε, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Οι Προδίνουμε συστάσεις και τεχνογνωσία για θέματα θαλασσίων μεταφορών. Επί τη βάση αιτήσεων από κράτη-μέλη επίσημους φορείς δίδουν δίδει αυτές τις αιτήσει στην Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών και ξεκινάει τη διαδικασία ανάβλωσης των μέσων αυτών. Παρακολουθεί τα αναβλωθέντα αυτά μέσα, κάνει μια έρευνα αγορά σε σχέση με τις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές για να μπορεί να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση και η ναύλωση αυτών των μέσων σε ανταγωνιστικές τιμές και δίδει και αξιωματικού σύνδεση με τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια τέτοιων ενεργειών στρατηγικών θαλασσίων μεταφορών. Το κέντρο αυτό είναι σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να δεχθεί και να επεξεργαστεί οποιαδήποτε αίτηση για θαλάσσιες στρατηγικές μεταφορές. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν και τους διεθνείς φορούς, φορείς που έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει. Η Ιταλία ήταν το πρώτο έθνος το οποίο συμμετέσχε στο AMSCC και σε χρονολογική σειρά ακολούθησαν οι εξής χώρες σαν μέλη του φορέα αυτού η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ολλανδία, η Πολωνία, συγγνώμη, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Και το Σεπτέμβριο 2010 και η Πορτογαλία. Και επιπλέον, όπως βλέπετε, το ΝΑΤΟ, ΣΕΙΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση Αθήνα έχουν υπογράψει συμφωνίες με το AMSCC στον τομέα των στρατηγικών θαλασσίων μεταφορών. Έχω, κάπου έχουν χαθεί δύο διαφάνειες. Πώς μπορεί ένα μέλος, πώς μπορεί ένα κράτος να γίνει μέλος του AMSCC. Καταρχήν, το κράτος ή ο φορέα θα πρέπει να υποβάλουν μια επίσημη αίτηση όπου θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να γίνουν μέλη του κέντρου αυτού. Θα πρέπει να είναι σαφέ ότι η αίτηση αυτή δεν σημαίνει υποχρέωση να υπάρξει τελική συμφωνία. Με την υποβολή αυτής τη επίσημης αίτηση ξεκινάει μια διαδικασία αξιολογήσεως από την ελληνική πλευρά και μια σειρά συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, τον οποίων ο στόχο είναι να καταλήξουμε σε ένα μνημόνιο κατανόηση και έγγραφα τεχνικών ρυθμίσεων βάσει των συμφερόντων και των δύο συμβαλωμένων πλευρών. Με την υπογραφή τη Τελική συμφωνία ξεκινάει η διαδικασία κύρωση και θέση σε εφαρμογή βάσει τη εθνική νομοθεσία. Προτού φτάσω στις ε, πρόσφατες εξελίξεις, Θέλω να αναφέρω κάποιες αποστολές που έχει φέρει σε πέρα στο AMSCC τα προηγούμενα χρόνια. Συγγνώμη που δεν έχω δυστυχώς τις διαφάνειες. Χρησιμοποιώντας την ικανότητα διάσωσης, έστειλε το MCC μηνύματα για την ενημέρωση πλοίων τα οποία βρισκόντουσαν σε περιοχές ε, καταστροφών. Στην περίπτωση του τσουνάμι, η τα πλοία αυτά απήντησαν μέσα σε 24 ώρες, ενώ στην περίπτωση του τυφώνα Κατρίνα, πέντε πλοία απήντησαν μέσα, σε δύο ώρες. Στην περίπτωση του Ιράκ υπήρξε η υποστήριξη 80, της μεταφοράς θαλασσίως από 80 τάγκς που ήρθαν από την Σλοβενία προς το Ιράκ και επίσης από τη Σούδα στην Ελλάδα στο, στο Κουβέιτ. Δώσαμε επίσης υποστήριξη για την, ε, τη Γαλλία. Το 2008 μετά από την ε, λήξη διαδικασίας υποβολής προσφορών υπήρξε η ε, υποστήριξη της δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τσάντ από το λιμάνι της Δουάλα στο Καμερούν. 2009 το κέντρο ε, εξεπλήρωσε πλήρως τη μεταφορά εξοπλισμού με θαλάσσια μέσα ε, χωρών που δεν θέλησαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες ακολουθώντας το μνημόνιο κατανόησης το οποίο είχαν, είχαν υπογράψει. Το MSCC δίνει και μόνιμη υποστήριξη στη δύναμη αντιμετώπισης κρίσεων του, ανθρωπιστικών κρίσεων του ΟΗΕ για τη μεταφορά υλικού το οποίο αποσκοπεί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Τέλος τον Ιούνιο του 2010 το AMSCC, ε, μετά από αίτηση του γαλλικού ναυτικού, υποστήριξε την άσκηση Emerald 2002-2010 που έλαβε χώρα το 2010. Επρόκειτο για την ε, ε, θέση σε χρήση πλοίων του εμπορικού ναυτικού στην περιοχή του, της Σενεγάλης για να υποστηρίξουν την συνολική αυτή επιχείρηση Emerald 2010. Βλέπετε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις στα πλαίσια του AMSCC 2022, μαζί με προσώπους του Ευρωπαϊκού Φορέα ε, ε, Άμυνας συζητήθηκαν οι πάγιες διαδικασίες, επιχειρησιακές διαδικασίες και επίσης η πλατφόρμα για την επιμελητιακή υποστήριξη της του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας. Ακολούθησε επίσης ένα συμπόσιο σε σχέση με την πλατφόρμα άμυνας υπό την υποστήριξη του ελληνικού φορέα για τα θέματα αυτά και με την υποστήριξη του ελληνικού ε, φορέα για την ναυτιλία και του φορέα των Ελλήνων εφοπλιστών. Τον Ιούλιο του 2010 έλαβε χώρα υπογραφή μια τεχνική ρύθμιση, η οποία αφορούσε την ελληνοϊταλική συνεργασία στον τομέα των στρατηγικών θαλασσίων μεταφορών. Και πιο πρόσφατα, όπως είπα προηγουμένω, στο τέλο του 2010, το Υπουργείο Άμυνα τη Πορτογαλίας υπέγραψε τα αντίστοιχα έγγραφα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το κέντρο αυτό. Η διαδικασία ε, υπογραφής και κύρωση τη ελληνοπορτογαλική συνεργασία για τι θαλάσσιες μεταφορέ είναι εν εξελίξη. Και εδώ σας δείχνω τα ζητήματα τα οποία είναι εν εξελίξη. Έχουμε το θέμα της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνας με στόχο <clears throat> να περιληφθεί στην πλατφόρμα ε, επιμελητιακής υποστήριξης από τρίτους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνάψουν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με το IMSCC. Τον Νοέμβριο του 2010 η Κροατία υπέβαλε μια επίσημη αίτηση να ενταχθεί στο κέντρο αυτό και να χρησιμοποιήσει οι υπηρεσίες του. Το κέντρο έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία ε, αξιολόγησης για το νέο αυτό μέλος. Βάσει της απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος από το 2008 έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία αναδιοργάνωση του κέντρου, το οποίο θέλει να αποκτήσει πολυτροπική μορφή συνδυάζοντας ικανότητες θαλάσσιων μεταφορών, εναέριων αερομεταφορών μάλλον και άλλων μορφών ε, μεταφοράς. Επίσης, η δεξαμενή πλοίων, η βάση δεδομένων για τη δεξαμενή πλοίων, όπως αναφέρεται. Αυτή η βάση δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική για το κέντρο μας. Το να έχει στην διάθεσή του μια βάση δεδομένων για πλοία, μεταξύ των οποίων πλοία του εμπορικού ναυτικού διαφόρων τύπων, τα οποία μπορούν να είναι διαθέσιμα για ενέργειες και επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την αποστολή του AMSCC. Η βάση αυτή δεδομένων επικαιροποιείται ετησίω από ναυτιλιακέ εταιρείε, οι οποίε με επιστολέ προθέσεων έχουν δηλώσει την πρόθεσή του να δίδουν πλοία στο AMSCC όταν υπάρχει αίτηση από τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια μια συμφωνία μη δεσμευτικού χαρακτήρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ποια είναι τα πλοία αυτά. Αυτή είναι η... Έχουν προσθεθεί επίσης άλλα 15 πλοία, οπότε συνολικά έχουμε περίπου 197 πλοία διαφόρων τύπων. Μετά από συζητήσεις με το Φορέα και την Επιτροπή Οκεανοπόρου, Οκεανοπόρων Ναυτικών Μεταφορών υπάρχουν και πλοία τα οποία υποστηρίζουν πλοία τα οποία έχουν ικανότητα κατάψυξης για να μπορούν να υποστηρίζουν και μελλοντικέ ενέργειες και επιχειρήσεις θαλασσίων μεταφορών. Το AMSCC έχει ήδη προβλέψει ορισμένε μελλοντικέ εξελίξεις. Καταρχήν, το να υπάρχει συνεργασία με ε, με μη στρατιωτικές εταιρείε σε σχέση με τις μορφές επικοινωνίας, το να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η αυτονομία βάσει του ISO 9001-2008, επέκταση των, του αριθμού των μελών του AMSCC και επίσης για να προωθηθεί ο πολυεθνικός του ρόλος που προωθεί την ευκαμψία και την αποδοτικότητα Προφανώς δεχόμαστε με μεγάλη ευχαρίστηση την υποστήριξη από άλλα κράτη-μέλη με χρηματικές συνεισφορές. Τέλος, μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε περισσότερη τεχνολογία μας σε σχέση με την παρακολούθηση νεναυλωμένων πλοίων. Θέλω να σας περιθυμίσω ότι όλες οι υπηρεσίες του AMS-CC δίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη του δωρεάν, διότι οι λειτουργικές δραστηριότητες το κόστος τους καλύπτεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος. Εδώ κλείνω λοιπόν την παρουσίασή μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και με στη διάθεσή σας για ενδεχόμενα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι θα σας υποβάλουν ερωτήσεις. Θα παρακαλέσω τώρα τον ε, ταξιέρχο Ρουσό να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Uh, uh, Γεια σα. Είμαι διοικητή, λοιπόν, ταξίαρχο ε, Ρουσό στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορών. Δεν θα διαβάσω τι ε, τις ε, διαφάνειες που έχουμε εδώ, αλλά θα τις σχολιάσουμε. Εδώ βλέπετε μια νέα διοίκηση γιατί δημιουργήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2010. Είναι πράγματι νέα. Αν δει κανείς ε, γενικότερα αυτή την διοίκηση και δείτε τους στόχους της, πρέπει να καταλάβετε ότι η νέα διοίκηση αυτή είναι κάτι το μοναδικό. Γιατί? Γιατί είναι η πρώτη φορά που ε, τέσσερα κράτη, και θα επανέλθω σε ποια είναι αυτά τα τέσσερα κράτη, αποφάσισαν να δώσουν τον λειτουργικό έλεγχο κατά τη διάρκεια περίοδου ειρήνης σε μόνιμη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε συγκεκριμένες αποστολές όπως το Κωσυφό πέδιο στο Αφγανιστάν κτλ. Αλλά σε περίπτωση περίοδου ειρήνης γενικότερα είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και δείχνει πώς μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων. Προφανώς θα μπορούσατε να πείτε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καινούριο, γιατί από την αρχή οι αερομεταφορές των διαφόρων χωρών ε, συνεργάστηκαν και έχουμε πολλά παραδείγματα με το Βερολίνο 48-49, το Σεράγεβο 92-96 και την εμπλοκή των αερομεταφορών και ε, των στρατιωτικών δυνάμεων και των ειρηνευτικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού μέσω των αεροπορικών δυνάμεων των διαφόρων χωρών. Πάντως τα μαθήματα από όλα αυτά ήταν ότι απαιτείται περισσότερη αποτελεσματικότητα και ο μοναδικός τρόπος ήταν η περαιτέρω ολοκλήρωση. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι να υπάρξει ένα ποιοτικό άλμα πέραν από την απλή συνεργασία. Προφανώς υπάρχουν και περαιτέρω προϋποθέσεις που οδηγούν τις χώρες όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία να προχωρήσουν σε αυτήν την ευρωπαϊκή διοίκηση. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει και σε επίπεδο δημοσιονομικό, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι η αεροπορική αυτή διοίκηση είναι πολυεθνική. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, δεν είναι ΝΑΤΟ, αλλά και οι δύο αυτές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το αρχηγείο αυτό, είναι διαθέσιμο για τις αποστολές όλων αυτών των διοικήσεων και των χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όπως βλέπετε σε αυτή τη συγκεκριμένη διαφάνεια, αυτή η αεροπορική διοίκηση είναι συμβατή και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010, όπως επίσης και με τα επίπεδα προσδοκιών και επίτευξης αποτελεσμάτων του ΝΑΤΟ του 2009. Ήδη από το 1989 ξεκίνησε η στρατιωτική συνεργασία που οδήγησε στην δημιουργία του στρατηγίου αυτού. Το Δεκέμβριο του 1999 υπεγράφει μια επιστολή για τις αερομεταφορές, τις αεροπορικές, συγγνώμη, στρατιωτικές μεταφορές μάλλον, και ε, βασικός στόχος εκείνη τη φάση ήταν ο συντονισμός. Ε, των ε, στρατιωτικών αυτών αερομεταφορών. Δημιουργήθηκε το 2004 το AESC, e, το Ευρωπαϊκό Κέντρο, υπήρξαν όμως ελλείψεις σε επίπεδο ε, προσωπικού και σε επίπεδο πολιτικής βούλησης. Γι' αυτό το 2006 υπεγράφει μια υποσχετική επιστολή από το Βέλγιο και την Γαλλία και τη Γερμανία συγγνώμη μετά ακολούθησε η Ολλανδία και το Βέλγιο και επίσης το 2007 υπεγράφει η ιδρυτική πράξη και το 2009 η εφαρμοστική διάταξη για τη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2010. Λοιπόν, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά κατά τομέα, τομεακά in organizations, difference in Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, εδώ συνθήκες σε κάθε χώρα και σε επίπεδο αεροπορικού στόλου και σε επίπεδο νοοτροπιών θα έλεγα και πολιτικής βούλησης ακόμα. Στην ουσία μέσω ενός εγγράφου ε, εκχωρείται ο λειτουργικός έλεγχος ορισμένων εναερίων μέσων και υπάρχει επίσης και ο λειτουργικός πυλώνας, λίγο πιο περίπλοκος, ο οποίος έχει σαν στόχο την εναρμόνιση των ε, διαδικασιών και των επιπέδων που ισχύουν για τις αερομεταφορές, την εκπαίδευση κτλ. Ε, του, τον, του προσωπικού του στόλου. Εδώ βλέπετε ποια είναι αυτά τα μέσα, που βρίσκονται στις χώρες μας και πού είναι όλες αυτές οι μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Στρατηγείο και οι οποίες ελέγχονται από το ATC, ε, Transport Cooperation. Αν θέλετε εδώ μπορείτε να δείτε τα είδη των αεροσκαφών, των εναερίων μέσων που είναι διαθέσιμα. Θα δείτε εδώ ποιοι είναι οι τέσσερις αεροπορικοί στόλοι και στο τέλος του 2011 θα έχουμε 165 ενέργεια μέσα στη διάθεσή μας. Μέχρι τώρα έχουμε ε, εκχωρητήρια από τρεις χώρες, από την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, το Βέλγιο θα ακολουθήσει. Ο στόλος που ελέγχεται από το ATC του Eindhoven βλέπετε ποιος είναι και ποια είναι τα ενέργεια μέσα. Είναι αρκετά περίπλοκο εδώ όπως βλέπετε αυτή η διαφάνεια να σας εξηγήσω πώς ελέγχονται τα μέσα του ATC. Τα κράτη ζητούν θα έλεγα μέσα για μεταφορά, αυτό είναι μια αίτηση κάνουν προς το ATC. Το ATC συγκεντρώνει τα αεροσκάφη τα οποία είναι διαθέσιμα και τα κατανέμει στις αιτήσει που υπάρχουν για τη χρήση τους. Τα κράτη δεν είναι αυτά τα οποία ελέγχουν πλέον τη χρήση των αεροσκαφών, αλλά είναι αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του ATC. Μέχρι τώρα η αρχική επιχειρησιακή μας ικανότητα θα πρέπει να αποτελείται από 11 επιμέρους κέντρα και θα έχουμε περίπου συνολικά προσωπικό που θα ανέρχεται σε 150 περίπου άτομα. Και βλέπετε εδώ ποιοι είναι οι σχηματισμοί του ATC κατά τη διάρκεια περίοδου ειρήνης επαναλαμβάνω. Βλέπετε ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής είναι διετούς διάρκειας, ξεκινάμε με τον Γερμανό διοικητή και μετά θα ακολουθήσει Γάλλος, και βλέπετε επίσης ότι έχουμε και δύο ε, ε, υποδιαιρέσεις εδώ σε διοικητικό επίπεδο και την ευθύνη της κάθε υποδιαιρέσης την αναλαμβάνει κατ' εναλλαγή η Ολλανδία και το Βέλγιο. Το ATC είναι σχετικά νέο βέβαια, αλλά παρόλα αυτά ανήκει θα έλεγα σε ένα τοπίο στρατιωτικής συνεργασίας προϋπάρχων Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε διαφορετικού τύπου σχέσεις με πάρα πολλές οργανώσεις και, ε, οργανώσεις ε, και ε, σχηματισμούς σε όλο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η Πολιεθνική Επιτροπή ε, και αποτελείται από τέσσερα με από τον πρόεδρο και από τον διοικητή συγγνώμη και το τέσσερα μέλη από κάθε χώρα. Και αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. και μέσω του EDA και μέσω του ATF. Θα μιλήσουμε για τον αεροπορικό στόλο, ε, τον ομόλογο αεροπορικό στόλο. Συνεργαζόμαστε βέβαια με τον στόλο αυτό. of studies and reports about building the so it's part of one of the of Υπάρχει επίσης και το MCC, το οποίο έχει έδρα και αυτό στο Eindhoven της Ολλανδίας, είναι καλύτερο εκεί και συνεργαζόμαστε εύκολα. Γιατί συνεργαζόμαστε εύκολα και υπάρχουν και δύο τα στα οποία συμμετέχουμε. Είναι ο, ο Ευρωπαϊκός Στόλος και υπάρχει κι άλλο ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υποσυζήτηση και μπορεί να υπογραφεί την άνοιξη του 2011 για το λεγόμενο European Air Group. Βλέπουμε εδώ ότι το γερμανικό σχέδιο υπευλήθη στις 15 Οκτωβρίου, μετά ακολουθήθηκε από το γαλλικό και το ε, ολλανδικό και ελέγχει το κέντρο πλέον το αεροσκάφη αυτά τα οποία δεν ελέγχονται πλέον από τις εθνικές διοικήσεις. Περιμένουμε τώρα τη μεταφορά, την εκχώρηση μάλλον αρμοδιότητας από το Βέλγιο. Δεν έχει έρθει ακόμα και μόλις ε, έρθει τότε οι σχηματισμοί θα είναι λειτουργικοί. Στις αρχές του 2011 και θα συνεχιστεί πλέον ο έλεγχος, η εποπτεία των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων των σχηματισμών μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν προκλήσεις, είναι καινοτόμο το σχέδιο αυτό το οποίο ακολουθούμε, ιδιαίτερα σε επίπεδο με τις τομεακές εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων από πλευρά των κρατών μελών. Υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία διατίθενται και αντίστοιχα είναι και πάρα πολλές οι ευθύνε και υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος. Το ATC θα πρέπει να γίνει αντικείμενο αναγνώρισης όχι μόνο από τη διεθνή κοινότητα αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη των κρατών μελών. γιατί σίγουρα προέρχεται από χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πάντα ένα σύστημα πληροφορικής, ε, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό από όλους τους σχηματισμούς και ήδη από τις αρχές του 2011 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα γενικότερα σε επίπεδο ηλεκτρονικής επικοινωνίας κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό και θα, γιατί θα διασφαλίζει την εναρμόνιση της χρήσης των μέσων αυτών. Πέρα από τις τεχνικές συμφωνίες απαιτείται μια νομική βάση, απαιτείται μια συνθήκη αν θέλετε, σχετικά με τις δυνατότητες που θα έχουν οι σχηματισμοί αυτοί να λειτουργούν στα πλαίσια μιας πολιτικής, σε ένα πολιτικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν θέματα επίσης κοινοτικά ή κοινωνική συγγνώμη, διάσταση, όπως επίσης και η σχέση με την πολιτική ε, της διεύρυνσης, να δούμε αν οι νέες χώρες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος σε αυτήν την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ελπίζω να ακολουθήσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, οπότε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τώρα την άποψη του ΝΑΤΟ ο κύριος Μπρούνο Κατίν, υπεύθυνο υλικοτεχνικής υποδομής. Ε, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de... Καλή σας ε, μέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην Ευρωβουλή για να κάνω την παρουσίαση αυτή για το ΝΑΤΟ σχετικά με την ε, στρατηγική, στρατηγικές αερομεταφορές. Πριν να προχωρήσω στην παρουσίασή μου θα ήθελα πρώτα να πω ότι μέσα στα πλαίσια ε, των στρατηγικών αερομεταφορών περιλαμβανομένουμε και ναυτικές και χερσαίες μεταφορές. Συνεχίζω στα αγγλικά. Θα ρίξω μια ματιά σήμερα μαζί σας πώς συνδυάζονται από τον ΝΑΤΟ οι μεταφορές σε αυτό το σημαντικό τομέα και τις ικανότητες της στρατηγικών μεταφορών από και προς αερολιμένες και λιμένες με συντονισμένο τρόπο. Για να μην μακρηγορήσω, θα προχωρήσω σύντομα στην ολοκλήρωση παρουσίασή μου και θα ακούσω μετά ερωτήσεις εάν συμφωνείτε. Πρώτα λοιπόν, ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στη στρατηγική του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνει ένα ορμαλείο πλαίσιο πολιτικής και δόγματος. Έχουμε έγγραφο πολιτικής που υποστηρίζει το δόγμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πρόκειται για το έγγραφο Στατιωτικής Επιτροπής 0336 κάθετος 3 και εκεί περιλαμβάνεται η στρατηγική αερομεταφορά η ευθύνη των χωρών μελών είναι κοινή για την ανάπτυξη, οργάνωση των ε, ικανοτήτων στατικών αερομεταφορών. Ωστόσο, το, το ΝΑΤΟ έχει την ύπατη ευθύνη για την ανάπτυξη και ε, διατήρηση των δυνάμεων ή των εθνικών τομέων τους, τμήματων τους. Επομένως και πολυμερών συμφωνιών με άλλες χώρες για να ε, έχει πρόσβαση σε πόρους είτε σε αγορές για την κτήση των πόρων αυτών. Το ΝΑΤΟ και οι χώρες του προσφέρουν τις ικανότητες αυτές και σε άλλους οργανισμούς για να βελτιστοποιηθούν οι τρόποι χρήσεως των ε, μέσων αυτών και θα αναφερθώ σε αυτούς τους οργανισμούς μετά που θα πρέπει βέβαια να ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες ε, του ΝΑΤΟ και να συντονίζονται στο ορθό επίπεδο. Το ΝΑΤΟ επίσης εκτελεί και έλεγχο κινήσεων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, έλεγχο του ενεργείου χώρου καθώς και των λιμανιών σήμερα στο Αφγανιστάν. Και των αερολιμένων δηλαδή στο Αφγανιστάν. Με μονάδα, πολυεθνική ομάδα συντονισμού. Άλλος τομέας όπου θέλουμε να υπάρξει τυποποίηση είναι η υποστήριξη πέραν των εθνικών συνόρων στον ενέργειο χώρο και πέραν των ε, χερσιών συνόρων. Για, για τις μεταφορές transit στον συστηματικό αυτό τομέα. Τώρα ας περάσω στην, στον συντονισμό. Ο συντονισμός γίνεται από το Συμμαχικό Κέντρο Συντονισμού Κίνησης στην Βελική Μόνς, που είναι υπεύθυνο απέναντι, ε, υπόλογο μάλλον, στον ε, ε, ανώτατο Ευρωπαίο Συμμαχικό Διοικητή και παίζει κρίσιμο ρόλο για την υποστήριξη, παράδειγμα, των επιχειρήσεων ISAF στο Αφγανιστάν με διαχείριση όλου του συντονισμού των χρονοθυρίδων, πτήσεων κλπ. Το EMCC συνεργάζεται και με το EUMS και το EUTC όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μου. Ακούσαμε ήδη για δύο άλλους, άλλες προσπάθειες συντονισμού, AMCC και η Δεν θα πω λοιπόν τίποτε άλλο για τις πρωτοβουλίες αυτές, παρά μόνο ότι θεωρούμε ότι είναι ευεργετικές στην πολυεθνική μας προσπάθεια και ότι πολλαπλασιάζουν έτσι το αποτέλεσμα των δυνάμεών μας. Το 1999 στην διάσκεψη κορυφής ε, της Ουάσιγκτον, το EMCCE, άρχισε την ζωή του ως ε, συντονισμός αφενός των ε, θαλασσίων μεταφορών και, αφενό, και αφετέρου των αερομεταφορών και μαζί επετέλεσαν το EMCCE με βάση το Ολλανδικό Eindhoven. Η επιτυχία του κέντρου αυτού είναι καλά θεμελιωμένη από την αρχή και τώρα έχει 23 χώρες μέλη που συμμετέχουν. Και υπάρχουν και ε, χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται όπως η Νέα Ζηλανδία και η Ουκρανία να συμμετάσχουν. Το συμμαχικό κέντρο συντονισμού δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Συνεργάζεται ωστόσο στενά με το AMCC, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των κινήσεων και μεταφορών μέσων του ΝΑΤΟ. Το AMCC δρά σε ε, ε, στρατηγικό επίπεδο, ενώ το AMCC στο ε, επιθυσιακό επίπεδο. Είναι σημαντικό για το, για το ΝΑΤΟ, το MCC και το SCC υποστηρίζουν το ISAF. Το e UMS έχει παρόμοιες ρυθμίσεις με όπως το MCC, όπως και το ΝΑΤΟ δηλαδή. Τώρα καθαρά για την πλευρά των ικανοτήτων που προέρχεται από, δια, από συντονισμό διαφόρων μέσων. Όπως θα αναμένατε, οι χώρες μέλη προσφέρουν βασικά τις ικανότητες μέσω εθνικών προμηθειών. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη να μεταφέρει και ε, τα δικά του μέσα, υλικό και προσωπικό, τηλεπικοινωνίες κλπ. Όλα αυτά βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνη, σε διαρκή συναγερμό και το ΝΑΤΟ επαφίεται στις χώρες μέλη για να προσφέρουν μέσα μεταφοράς σε ε, δεν προτίθεμαι να καλύψω όλες τις ικανότητες που ήδη εξηγήθηκαν. Θα περιοριστώ λοιπόν μονάχα στις ικανότητες, στην πρωτοβουλία ικανότητας ε, ε, στατικών αερομεταφορών, την ΝΑΜΣΑ. Θα έλθω επίσης και στις στατικές θαλάσσιες μεταφορές, που επίσης είναι κρίσιμες για τον ΝΑΤΟ. Συχνά λησμονούν οι ε, άνθρωποι ότι υπάρχει, υπάρχουν και οι θαλάσσιες μεταφορές που είναι σημαντικός πολλαπλασιαστής της δυνάμεως μιας συμμαχίας και είναι πολύ πιο οικονομικές εάν υπάρχει επαρκής χρόνος. Η ικανότητα στρατηγικής μεταφοράς του ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους μέσα από μια κοινή ε, συνεργασία. και ιδίως με την κτήση αεροσκαφών που είναι ικανά να μεταφέρουν μεγάλα φορτία. Ήδη από το 2006 δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία για την αγορά αεροσκαφών σε 17. Ήδη έχουμε τώρα στη, στην βάση στην ε, Ουγγαρία με αεροσκάφη σε 17. Έχουμε και την ΝΕΜΑ επίσης NAMA Airlift Agency που επίσης έχει αεροσκάφη C-17 του ΣΑΚ, του προγράμματος ΣΑΚ. Ασφαλώς στη σύντομη ιστορία της η πτέρυγα έχει ε, σημαντικές επιχειρήσεις στο ενεργητικό της, όπως βλέπετε στην ε, διαφάνεια αυτή. Και κυρίως βέβαια στην υποστήριξη της επιχειρήσης ISAF. Η ΣΑΚ παραμένει ανοιχτή στη συμμετοχή και άλλων χωρών εφόσον αυτό απαιτηθεί. Στον χώρο αυτό επίσης η πτέρυγα αερομεταφορών μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον και άλλα αεροσκάφη εκτός από τα και αυτά. Σε ό,τι αφορά την ΝΑΜΣΑ τώρα, δηλαδή ε, είναι ο οργανισμός του ΝΑΤΟ που είναι αρμόδιος για ε, συντήρηση και έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Επίσης στενή συνεργασία με την βιομηχανία και έχει διαρκείς συμβάσεις για την χρήση των διαφόρων μέσων σε μεγάλη ταχύτητα. Προσφέρει επίσης διοικητική υποστήριξη στην ΝΑΜΑ και διαχειρίζεται την τη σύμβαση Σάλης. Όπως σας είπα πριν, η Σάλης, στην οποία συμμετέχει η Νάμσα, είναι κυρίως η διαχείριση της συμβάσεως με 18 χώρες που συμμετέχουν ήδη στην Σάλης και που λύγει το Δεκέμβριο του 2010 η σύμβαση αυτή, αλλά τώρα ανανεώνεται για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε δύο Αντόνοφ ε, έτοιμα να απογειωθούν όταν χρειαστεί και άλλα δύο τα οποία ε, μπορούν να κινητοποιηθούν μέσα σε προθεσμία έξι ημερών. Και οι χώρες έχουν συμφωνήσει τώρα να ε, συμβάλλουν με 2.500 ώρες πτήσης τον χρόνο. Όπως είπα πριν, η τρέχουσα σύμβαση λίγη τον Δεκέμβριο του 2010 και η Νάμσα διαπραγματεύεται τώρα την ανανέωσή της μέχρι τέλη του 2012. Εάν συνεχίσει να υπάρχει καθυστέρηση στα δικά μας προγράμματα, η ενδιάμεση λύση που είναι η Σάλης θα χρειαστεί ίσως να συνεχίσει να λειτουργεί και περισσότερο από όσο έχουμε μέχρι τώρα σχεδιάσει. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, γιατί είπα πριν ότι αυτές είναι συμπληρωματικές. Η Συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή, έχει εντοπίσει ότι υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα στις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές. Και αναμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και βασισμένο στη νέα στρατηγική αντίληψη για το 2012. Για να διαχειριστούν καλύτερα τα μέσα της, ε, των θαλάσσιων μεταφορών. Έχουν φτιάξει οι χώρες ε, του ΝΑΤΟ την ε, Διευθυντική Επιτροπή με συμμετοχή 10 χωρών και προσκαλούνται και άλλες χώρες για να συμμετάσχουν. Αυτή η Διευθυντική Επιτροπή, η Διαχειριστική Επιτροπή διαχειρίζεται διαφορετικές συμβάσεις που ε, γίνονται με μία εταιρεία η οποία προσφέρει σκάφη τα λεγόμενα ρόρο και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δικές του, δικές του ικανότητες ικανότητες θαλάσσιων μεταφορών που διαθέτει και στις ε, άλλες χώρες μέλη. Υπάρχουν και άλλες ικανότητες που διατίθεται μέσω αυτής της ε, πρωτοβουλίας, όπως για παράδειγμα της Δανίας, που ε, αύξησε τις ικανότητες αυτές, καθώς και τη Γερμανία που ε, μπήκε από πέρσι. και να αναπτυχθούν οι ικανότητες της SEC με την συμπερίληψη και άλλων χωρών. Όπως είπα, το πλαίσιο της, ε, του δόγματος είναι ρωμαλαίο. Ήδη από το 1999 όπου διαπιστώθηκαν οι ανάγκες αυτές. Ωστόσο δεν έχουμε με σταυρωμένα τα χέρια, διαπιστώνουμε που βρίσκονται οι ελλείψεις που αυτές είναι δυνατόν να τις διαχειριστούμε με ε, πρωτοβουλίες. Πολλοί Πολυάριθμα αριθμα προγράμματα, πολυεθνικά προγράμματα ε, ε, εξασφαλισμένης πρόσβασης έχουν προσφέρει σημαντικές ικανότητες και έχουν, παίζουν κρίσιμο ρόλο ως πολλαπλασιαστής δυνάμεως. Το ΝΑΤΟ έχει επιμείνει και έχει προωθήσει πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές, ωστόσο οι περισσότερες έχουν αναλυθεί από τις ίδιες τις χώρες. Ε, τα δύο βασικά πολυεθνικά κέντρα συντονισμού είναι υπόλογα στη, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνεργασία και η εκπαίδευση παραμένουν ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ. Και έγινε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση αυτά στην τελευταία διάσκεψη κορυφή στην Λισαβόνα. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικέ ελλείψει ε, στι στατικέ θαλάσσιε ικανότητε μεταφορά. Και αυτέ πρέπει να αντιμετωπιστούν. Λίγη εδώ η παρουσίασή μου και περιμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε όλες τις παρουσιάσεις για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα και να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον στρατηγό Βιντσέντσο Πούρη να κάνει τη δική του παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να αναφερθώ στο ρόλο του στρατηγικού προσωπικού του ΝΑΤΟ για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις θαλασσίων μεταφορών. <clears throat> Καταρχήν, θα ήθελα να σας, να σας εξηγήσω ποια είναι η θέση μου. Εγώ είμαι ο υπεύθυνο υλικοτεχνικής υποστήριξης επιμελητίες, δηλαδή του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω ένα επιτελείο από 30 περίπου άτομα που υποστηρίζει από την 1η Ιανουαρίου θα μεταφερθεί στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες σε διάφορες πτυχές της υλικοτεχνικής υποστηρίξης, κίνηση και μεταφορές ιδίως αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές, συντονισμό, υποστήριξη συντονισμού, ε, ιατρικές και άλλες υπηρεσίες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει στη διάθεσή του ιδιόκτητα αεροσκάφη. Δεν υπάρχει μόνιμη αεροπορική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό εξαρτώμεθα απόλυτα από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στις αποστολές μας και περιμένουμε να ανταποκρίνονται στις αιτήσει μας υπήρξε μια σύμφωνη από το 2006 να μπορεί το, η, ο, η, η υπηρεσία υλικοτεχνικής υποστήριξης να υποστηρίζει δράσεις, παραδείγματος χάρη, του ανθρωπιστικού φορέα ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τμήματος που έχει να κάνει με τις πληροφορίες και τις μετακινήσεις του ΜΙΚ. Δημιουργήθηκε μέσα στο UMS μια ιδιαίτερη υπηρεσία για να υποστηρίξει τέτοιου είδους ενέργειες. Ο μηχανισμός αυτός ετέθη πρώτη φορά σε λειτουργία το 2006 όταν έδωσε στρατηγική αερομεταφορά ε, για αντιμετώπιση πλημμυρών στην Αλγερία. Η χρήση λοιπόν μέσων πολιτικού χαρακτήρα και στρατιωτικού ε, χαρακτήρα αναφέρει ότι για την ανακουφιστική δράση οι στρατιωτικές υποδομές είναι οι υποδομές τελευταίας καταφυγής. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει κανείς με μη στρατιωτικούς πόρους και μέσα να δημιουργήσει τι απαραίτητε τις απαραίτητες υποδομές στο χρονικό διάστημα που απαιτεί η Κομισιόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στρατιωτικές υποδομές και μέσα για να μπορέσετε να επιτύχετε το στόχο αυτό το ταχύτερο δυνατό. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι δεν έχουν ποτέ την ηγετική ε, ευθύνη οι στρατιωτικέ δυνάμει για ενέργειε ανθρωπιστική και ανακουφιστική βοήθεια, και είναι πάντα οι πολιτικέ αρχέ Και στη δική μα περίπτωση η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ Ανθρωπιστικών Δράσεων τη Κομισιόν. Ο στόχο μα είναι να έχουμε ταχεία αντίδραση και δράση, όχι μόνο στον τομέα τη στρατηγική αερομεταφορά ή ναυτική μεταφορά, αλλά και για κάθε μορφή υλικοτεχνική υποστήριξη. Όπω είπα στην αρχή, εμεί καλύπτουμε το πλήρε φάσμα υλικοτεχνικής υποστήριξης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επαφή με τα σημεία επαφής των κρατών μελών, με τους διεθνείς φορείς. Όταν λέω εθνικούς, ε, εθνικά σημεία επαφής, τις στρατιωτικές, τα στρατιωτικά σημεία επαφής με διεθνείς φορείς και υπηρεσίες που μας επιτρέπει να ζητήσουμε κάθε μορφή υλικοτεχνικής υποστήριξης. Αυτό έγινε πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στο Πακιστάν. Στις 18 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά από τις πλημμύρες του Πακιστάν, το ΜΙΚ ζήτησε επίσημα την υποστήριξη του UNPC για να μπορέσει να βοηθήσει στη μεταφορά ζωτικών ε, εφοδίων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Αυτά τα εφόδια είχαν τύχει υποσχέσεων από τα κράτη-μέλη και από μη κυβερνητικού φορείς. Μετά από συγκεκριμένες αιτήσει από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς του Πακιστάν. Η ομάδα σχεδίασης ήρθε σε επαφή με την υπηρεσία MMCE και άλλωστε στις πρωτεύουσες των κρατών μελών για να πάρει μέσα αερομεταφορών τα οποία μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για την ενέργεια αυτή. Τις επόμενες μέρες το ENPC λειτουργήσε ως διαδραστική επιφάνεια μεταξύ Τσεχίας, Φιλανδίας και των αντίστοιχων φορέων αεροπορικών μεταφορών και του ΜΙΚ από την άλλη πλευρά. Ως αποτέλεσμα αυτού του συντονισμού, τρεις τέτοιες πτήσεις έγιναν από την, στις αρχές Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Πακιστάν. Καταρχήν ένα, σκάφ, ένα αεροσκάφος Αντόνοφ 124, τσεχικού χαρακτήρα, τσεχικής ιδιοκτησίας που μετέφερε φορτία από την Ιταλία Μπρίντεζη και από τη Λιψία. Περίπου 100 τόνους μετέφερε στις 30 Σεπτεμβρίου στην Ισλάμ Αμπάντ. Η πτήση αυτή έγινε βάσει του συστήματος σάλις που ανέφερε προηγουμένως ο σα συναδελφός μου. Ένας δεύτερο, <coughs> μια δεύτερη πτήση με Αντόνοφ 124 πάλι από την εισαγική ε, Δημοκρατία ξεκίνησε από το αεροδρόμιο των East Midlands στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετέφερε 75 τόνους στο καράτσι από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Σεπτεμβρίου. Και πάλι επί τη βάση του συστήματος Σάλης. Τρίτη πτήση ενός αεροσκάφου C-17 στρατιωτικό αεροσκάφος της Φιλανδίας <clears throat> με 40 τόνους από, από τη Δανία, 40 τόνους οι οποίοι έφτασαν στις 16 Σεπτεμβρίου στην, ε, στο Καράτσι και έγινε αυτή η μεταφορά βάσει του συστήματος ΣΑΚ strategic airlift capability. Ένα, ένα τμήμα τη δεύτερη μεταφοράς πήγε στο Γκάλεν Κίρχεν στη Γερμανία και μετά από εκεί στο Πακιστάν με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Αυτό δείχνει λοιπόν και τη συνεργασία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φορέα μας και του ΝΑΤΟ. Στο δεύτερο μισό του Αυγούστου και το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου ήταν για μας μια περίοδος έντονου σχεδιασμού και επαφών για πολλούς φορείς. Το τελικό αποτέλεσμα όμως μπορεί να θεωρηθεί πάρα πολύ επιτυχές. Η συνολική αυτή αντιμετώπιση χρησιμοποιείται πάρα πολύ, η έκφραση μάλλον χρησιμοποιείται πολύ, αλλά μπορώ να σας πω ότι στη δική μας περίπτωση υπήρξε απόλυτη αντιμετώπιση σε συνολικό επίπεδο με συνεργασία και των κρατών μελών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και των στρατιωτικών επιτελείων όλων των κρατών μελών, πολλών κρατών και με εμπορικούς φορείς, που, ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι συμμετέσχαν. Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε. Έχουμε μάθει πολύ σημαντικά μαθήματα επί τη βάση επιτυχιών και όχι αποτυχιών. Αυτό το οποίο είναι σαφές από αυτή την ιδιαίτερα θετική εμπειρία είναι ότι η στρατιωτική συνιστόσα μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να υποστηρίξει δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακούφιση καταστροφών. Επί των κατευθυντήων γραμμών του Όσλο για τη χρήση πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για ανακουφιστικές ενέργειες. Ο τομέας στρατιωτικής, στρατηγικής αερομεταφοράς είναι ένας τομέας ο οποίος <clears throat> είναι σημαντικός περισσότερο στα κράτη-μέλη από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως τα μέσα των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως στρατηγικές αερομεταφορές μας δίνουν επίσης μεγάλη ευκαμψία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε διάφορες περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλές <clears throat> διευκολύνσεις για ε, λιμένες και αερολιμένες. Φυσικά και οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο όταν πρέπει να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες υλικού αλλά σε, σε μεταγενέστερες ε, ενέργειες ανακουφιστικού χαρακτήρα υποστηρίζοντας κυρίως αερομετοφερόμενες επιχειρήσεις. Από το Σεπτέμβριο το UNMIC, το MIC και το ENPC εξακολουθούν να συνεχίζουν τις διαδικασίες αυτές που προανέφερα και για τη μελλοντική συνεργασία και την, επίσης τις κοινέ ασκήσεις εκπαίδευσης όπως ε, ε προκύπτει και από το κοινό έγγραφο της Κομισιόν και των κρατών μελών 26 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι έχουμε ε, δημιουργήσει ένα έφορο πλαίσιο για συνεργασία μετά από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας για το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ στρατηγέ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Δημήτριος Μουτσιάκης από τη Διεύθυνση Υλικοτεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Θα ξεκινήσω αμέσως την παρουσίασή μου. Ο κατάλογος ε, προόδου του Ελσίνκη του 2003 δείχνει ποιες ήταν οι σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο στρατηγικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανεπίσημη συνάντηση του 2010 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων διευκρινίστηκε ότι οι απαιτήσει σε επίπεδο στρατηγικών μεταφορών είναι βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα τώρα με τους αρχικούς στόχους του 2010, υιοθετήθηκε ε, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και η Στρατηγική Συνεργασία των Πολεμικών Σχηματισμών και φάνηκε για μια ακόμη φορά μεγενθυμένη θα έλεγα η έλλειψη των αναγκών για, τις, ε, για αυτού του είδους τις μεταφορές. Η αρχική στόχη του 2010 αναφέρθηκαν επίσης στις βασικές ελλείψεις, στις κρίσιμες ελλείψεις που υπάρχουν ιδιαίτερα στις στρατηγικές αερομεταφορές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν αναλυφθεί πολλαπλές πρωτοβουλίες για να ελαφρυθεί το πρόβλημα στον τομέα των μεταφορών και αερομεταφορών και όλες αυτές αναφέρθηκαν και από τον συνάδελφο του ΝΑΤΟ και δεν θα τις ε, θέσω λεπτομερώς. Σε επίπεδο στρατηγικών αερομεταφορών υπήρξαν πρωτοβουλίες, υπήρξε επίσης και το Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο Συντονισμού και το ε, Ευρωπαϊκό Στρατηγείο. Βασική στόχη είναι ακριβώς να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των μέσων και η καλύτερη χρήση των μέσων, η πιο αποτελεσματική τους χρήση. Δεν θα αναφερθώ στις θαλάσσιες στρατηγικές μεταφορές. Ξέρουμε τι διαστάσεις υπάρχουν απόψεων ανάμεσα στα διάφορα <clears throat> στις ε, διάφορες θέσεις που έχει ο καθένας, αλλά δεν διαπιστώνεται πολύ μεγάλη έλλειψη και υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των εθνικών κέντρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την υπηρεσία το Μάιο του 2006 να κάνει μία ανάλυση σε βάθος, συνολική ανάλυση των μελογικών στρατηγικών αναγκών στον τομέα των αερομεταφορών, ιδιαίτερα για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ε, να κάνει τις απαιτούμενες συστάσεις η δική μου υπηρεσία. Για να το πετύχει αυτό, η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία λοιπόν ξεκίνησε τις μελέτες, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Ε, οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν χρήσιμα συμπεράσματα και χρήσιμες συστάσεις, οι οποίες ε, παρουσιάστηκαν εν μέρη και από το EDA, αλλά μια συνολική έκθεση με τη λεπτομερή ανάλυση όλων των ε, προαναφερθησών μελετών ε, θα υποβληθεί από πλευράς της, Εθνική, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής ε, Άμυνας στο τέλος του επομένου έτους και οι προσπάθειες που γίνονται τώρα είναι συμπληρωματικές με αυτές που είχαν γίνει παλαιότερα. Προσπαθούμε να βρούμε με ποιον τρόπο καινοτόμα μέσα θα μπορέσουν να επηρεάσουν τις στρατηγικές αερομεταφορές. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στον τομέα των αερομεταφορών που μας ενδιαφέρει το λεγόμενο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Στόλου Αερομεταφορών. Αναγνωρίστηκε ότι τα κράτη-μέλη θα εμπλακούν περισσότερο σε διαχείριση κρίσεων στο μέλλον και αναγνωρίζοντας επίσης ότι υπάρχουν περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αναπτύχθηκε ο ευρωπαϊκός αυτός μεταφορικός στόλος για να αναπτύξει τις ικανότητες και να καλύψει τις ανάγκες των εθνικών κέντρων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων πιθανώς διεθνών οργανισμών. Ε, αποφασίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 2008 η δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού με ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα το οποίο θα εξετάσει τα βιώσιμα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μεταγωγικού Στόλου. Στις 10 Νοεμβρίου του 2008 οι Υπουργοί Άμυνας 12 κρατών μελών υπέγραψαν μία δήλωση προθέσεων και ε, υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους για να καλύψουν τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Η αρχική ιδέα για, την ευρωπαϊκή, για τον ευρωπαϊκό αυτό στόλο ήταν ε, θα έλεγα γύρω από το αεροσκάφος Α400M βασικά. Είχε χτιστεί γύρω από το αεροσκάφος Α400M. Αλλά ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής τώρα έχει διευρυνθεί για να περιλάβει και άλλους τύπους αερομέσων λόγω ακριβώς και των καθιστορήσεων που παρατηρούνται στην παράδοση των πρώτων framework Λοιπόν, έτσι θα καλυφθούν τα θέματα ε, των αναγκών από διάφορους μηχανισμούς και διαφορετικούς σχηματισμούς, ιδιαίτερα γύρω από τα Α400M όταν τεθούν σε υπηρεσία. Μετά από την επιστολή προθέσεων του 2009 από τους 15 ε, Υπουργούς Άμυνας, απέδειξε η υπογραφή αυτή την ξεκάθαρη πολιτική βούληση για να προχωρήσουν στη ρύθμιση και στρατιωτικών θεμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά κράτη αναγνωρίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών βελτιωμένων και αποτελεσματικών μπορεί να βοηθήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ε, κατανομής ε, του διαμοιρασμού και της ε, απόκτησης από κοινού δυνατοτήτων είτε μέσων είτε εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε διαχείρισης εμπορευμάτων κτλ. Τον Μάρτιο του 2011 θα έχουμε την κατάληξη των νέων προγραμμάτων και θα ε, κατατεθεί επίσης και το νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός προγράμματος κατηγορίας Α που θα συνδυάζεται με επιμέρους προγράμματα κατηγορίας Β τα οποία θα συναποτελούν τις υποχρεώσεις αλλά και τη νομική βάση για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας. Το πρότυπο ATF, όπως βλέπετε εσείς, το ATF είναι μια εταιρική σχέση που έχει σαν στόχο την βελτίωση της παροχής και της αποτελεσματικότητας υπηρεσιών αερομεταφοράς μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου ανάμεσα στις συμμετέχουσες και πολιτικά θα έλεγα πρόθυμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μονάδες οντότητες που ασχολούνται με τις αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ένα εύκαμπτο πλαίσιο το οποίο δεν αποκλείει κανέναν και δεν αποκλείει τη συνεργασία ανάμεσα σε αθνικές και πολυεθνικές ε, μορφές ε, στόλου και επίσης έχει σαν στόχο τη χρήση όλων των μέσων και στο παρόν και στο μέλλον ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους ή προέλευσής του. Εμείς θέλουμε ένα δίκτυο στόλου AETF, τα οποία να είναι διαθέσιμα μέσω των συμμετεχουσών χωρών για την κάλυψη των στρατιωτικών τους αναγκών. Η βασική στόχη του προτύπου ATF e περιλαμβάνονται και στην επιστολή προθέσεων η οποία υπεγράφει από τους 15 Υπουργούς Άμυνας. Πρώτος στόχος και ο γενικότερος στόχος είναι η βελτίωση των αερομεταφορών στρατιωτικού τύπου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η ανάπτυξη καλύτερων μέσων για τη χρήση των υπαρχουσών και μελλοντικών δυνατοτήτων και η ανάπτυξη επίσης ε, ε, τρόπων βελτίωσης, μέσων βελτίωσης των δομών και οργανώσεων γύρω από τις στρατηγικές αερομεταφορές. Οι μέθοδοι εργασίας, τα επίπεδα συμμετοχής μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά παρόλα αυτά όλες αυτές οι προσπάθειες θα γίνονται αντικείμενο συντονισμού στο καταλληλότερο κάθε φορά επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή από τα κράτη-μέλη και από τις οργανώσεις των κρατών μελών που ασχολούνται με τις αερομεταφορές θα οδηγήσουν ακριβώς και τις δυνατότητες εθελοντικής συμμετοχής και κατά περίπτωση συμμετοχής στον στόλο AETF. Ε Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια συμπληρωματική δομή μεταφορών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχύσουμε την κάλυψη των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι σε ανταγωνισμό με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διοίκησης, Μεταφορών ή αδίποτε άλλη μορφή συνεργασίας. Θέλουμε όμως να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πρωτοβουλειών, θέλουμε να αποφύγουμε τις, αποκαλ... τις επικαλύψεις των προσπαθειών αυτών και για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται καλύτερη ενημέρωση και συνεργασία με όλες τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπετε στον γαλανό χώρο, στη γαλανή περιοχή, τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα των, της συνεργασίας της αεροπορικές μεταφορές. Φαίνεται περίπλοκο και δυσνόητο, αλλά δεν είναι. Από τις δύο πλευρές θα βλέπετε τις διάφορες δυνατότητες οι οποίες ε, είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την υπηρεσία. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να καλυφθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει λόγω της έλλειψης πόρων και του επίπεδου στήριξης από την πλευρά των κρατών μελών, των δημοσιονομικών περικοπών δηλαδή, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Πιο σημαντικός είναι ο κίτρινος τομέας, όπου μπορείτε να δείτε εδώ την ε, διαλειτουργική ε, σχέση για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Σχετικά τώρα με τις ε, ενεξελίξει επιχειρήσεις και στα πλαίσια του ATF έχουμε ξεκινήσει μέχρι τώρα τέσσερις μελέτες. Η δεύτερη και η τρίτη αυτή τη στιγμή εξελίσσονται. Πιο σημαντική είναι η μελέτη καθορισμού των στόχων και ε, η τελική διατύπωση της έκθεσης αυτής ε, κατατέθηκε πριν δύο μήνες και ήδη στις αρχές του χρόνου οργανώσαμε ένα, μια συζήτηση με συμμετοχή των κρατών μελών για να στοχεύσουμε στην τελική διατύπωση των ανακών και των σχηματισμών που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτές. Μια άλλη μελέτη είναι η μελέτη διπλωματικών διευκολύνσεων η οποία προσπαθεί να εναρμονίσει τους μηχανισμούς αυτούς τους διπλωματικούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο, ε, μια άλλη συζήτηση του 2011 θα έχει σαν στόχο εκ νέου την ανάλυση αυτού του ιδιαίτερα περίπλοκου θέματος και να καταστήσει ικανές τις ε, διοικήσεις να μπορέσουν να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ήδη υπάρχει συνεργασία στα θέματα τα οποία θεωρήθηκαν κατά προτεραιότητα σημαντικά από τα κράτη-μέλη. Το ένα θέμα είναι η διακυβέρνηση όλων αυτών των μηχανισμών, διακυβέρνηση δηλαδή του ATF και το νομικό του πλαίσιο. Δεύτερον είναι η συνεργασία σε επίπεδο λειτουργικό αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Ουσιαστικά είναι προσπάθειες εναρμονισμού εδώ. Και το τρίτο είναι η ομάδα εργασίας για τις λεγόμενες diplomatic clearances στην ουσία προσπαθούμε να εναρμονίσουμε και να απλουστεύσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους χορηγούνται αυτές οι διπλωματικές διευκολύνσεις. Πέραν αυτών των ομάδων εργασίας υπάρχουν άλλες έξι μέχρι τώρα ομάδες. Αλλά όπως σας είπα, λόγω ακριβώς της έλλειψης φόρων δεν έχουν ακόμα συσταθεί σχετικά με τις διπλωματικές αυτές διευκολύνσεις έχουν σαν στόχο την διασφάλιση της ε, ελεύθερης κίνησης των αεροσκαφών στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους απαιτήσεις και σχετικά με την υπέρπτυση μιας χώρας μέλους προκαλούν καθυστερήσεις και παρεμποδίζουν την ταχεία εκτέλεση των επιχειρήσεων. Αυτός ο μηχανισμός τύπου legacy θα πρέπει να αλλάξει. Single European Sky in the coming years. The relative co working group is developing under the of umbrella the legal framework Προτείνεται λοιπόν ένα πλαίσιο έτσι ώστε να υπάρξει ένας εναρμονισμένος μηχανισμός χορήγησης αυτών των διπλωματικών διευκολύνσεων αν θέλετε και ταυτόχρονα να υπάρχει μια ευρύτερη περιοχή για την οποία δεν θα εφαρμόζονται αυτές οι διπλωματικές ε, διευκολύνσεις. Περιμένουμε εν πάση περιπτώσει προτάσεις από πλευράς των κρατών μελών σε πολλούς από αυτούς τους τομείς Υπάρχουν θέματα που αφορούν τις χώρες μέλη λοιπόν, ιδιαίτερα στον τομέα των στρατιωτικών αεροσκαφών. Εφόσον ρυθμιστεί το θέμα αυτό θα γίνουν ικανά τα κράτη-μέλη να λειτουργούν στο ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο χωρίς να ζητούν πάντα να υπάρξει μια αδειοδότηση για κάθε μία ξεχωριστά από τις πτήσεις αυτές. Αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα την χρήση του διαθέσιμου εναερίου χώρου και υπάρχουν και αρκετά θέματα περιβαλλοντικά τα οποία τίθενται εδώ, πέραν των διοικητικών ρυθμίσεων. Το θέμα αυτών των διπλωματικών διευκολύνσεων είναι και διπλωματικό αλλά και θέμα πολιτικό βαθύτατα. Και γι' αυτό οι μηχανισμοί στους οποίους θα καταλήξουμε θα εξαρτηθούν κατά πολύ από την πολιτική βούληση για αλλαγή. Υπάρχουν τέσσερα θέματα τα οποία θα πρέπει βασικά να ρυθμιστούν πέραν της ε, γενικότερης στρατηγικής. Υπάρχει το θέμα των στρατιωτικών αεροσκαφών τα οποία επιχειρούν στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών συνόρων, μη ευρωπαϊκών αεροσκαφών τα οποία εισέρχονται στον εναέριο ευρωπαϊκό χώρο και τέλος η χρήση των εμπορικών αεροσκαφών, μεταγωγικών πάντα, για ε, στρατιωτικούς λόγους. Δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά το πρώτο που θα πρέπει να λυθεί είναι το θέμα της ελευθερίας κίνησης των λεγόμενων κρατικών αεροσκαφών. Βέβαια δεν υπάρχει κοινός ορισμός για το τι είναι ένα κρατικό αεροσκάφος μέχρι τώρα. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις γι' αυτό. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνεκτική στρατηγική σχετικά με τις διπλωματικές διευκολύνσεις. Εδώ μου λείπει ε, μια διαφάνεια. Uh, were better depicted in a, in a figure, in a figure like the ε, Λοιπόν, είναι περίπλοκο το θέμα εδώ, ιδιαίτερα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα βρίσκει λύση. Εμείς προτείνουμε 7 διαφορετικές ε, επιλογές έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα των διπλωματικών διευκολύνσεων. Ξεκινάμε με την απλούστευση των αιτήσεων και συνεχίζουμε μέχρι και την 7η επιλογή η οποία προβλέπει την δυνατότητα μιας μονάδας διπλωματικών διευκολύνσεων στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πριν αντιμετωπιστούν βέβαια τα θέματα τα οποία άπτονται της παρουσίας μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να λύσουμε τα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα για το εσωτερικό μας. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε την εφαρμογή πρώτα της επιλογής 1 και της επιλογής 5. Να απλουστεύσουμε δηλαδή τις αιτήσει και να δημιουργήσουμε ένα clearing board, ένα διαχειριστικό κέντρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή εκκρεμότητες ε, και που δεν έχουν κλείσει ουσιαστικά το θέμα της διακυβέρνησης του ATF και της νομικής μας βάσης και θα πρέπει να κλείσουμε και τις δύο μελέτες αυτές σχετικά με τις διπλωματικές διευκολύνσεις. Όπως επίσης και το θέμα της κοινή χρήσης των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το θέμα της δικτύωσης των στόλων, το θέμα των πολιεθνικών ε, μονάδων μεταφορών και το θέμα της αποκοινού απόκτησης αεροσκαφών. Θα ήθελα επίσης να μην καθυστερήσω πάρα πολύ στη συγκεκριμένη διαφάνεια, να πω ότι γίνεται σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ε, για τα Ελικόπτερα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο χρήσης των ελικοπτώρων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την αύξηση της διαθεσιμότητας των ελικοπτέρων. Αυτό ζητήθηκε και από πλευράς του ΝΑΤΟ. Γίνονται από εκεί προσπάθειες, προσπαθούμε και εμείς να υποστηρίξουμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Ήδη υπάρχουν κάποια βασικά βήματα από τότε που ξεκινήσαμε με τις δύο ασκήσεις κατέτος στη Γαλλία και στην Ισπανία με 50 ελικόπτερα και 1.300 άτομα προσωπικό. Ε, θέλουμε να προχωρήσουμε και με τη διοργάνωση δύο ακόμα ασκήσεων κατέτος, η μία να αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε περίπτωση κλιματολογικών αλλαγών υπερβολικά ζεστής θερμοκρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας ή στην ύπαρξη πάρα πολύ υψηλών επιπέδων κονιορτού. Έτσι θα διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα όλων αυτών των μέσων και θα πετύχουμε τους στόχους μας όπως το πολυεθνικό σμήνος ελικοπτέρων, τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε να βρεθούν κοινέ ευκολότερα λύσεις, να αξιολογήσουμε επίσης το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να βοηθήσουμε επίσης την ε, εκπαίδευση και την επιχειρησιακή χρήση ε, για την σωστή ε, ανάπτυξη των μονάδων ελικοπτέρων NH90 για να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί και τέλος είμαστε σε μια πολύ πρώιμη φάση εδώ βέβαια είμαστε ακόμα στο επίπεδο σχεδιασμού Πολλά από τα, πολλές από τις συμμετέχουσες χώρες μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση για εκπαιδευτικές ομάδες ε, κάλυψης των αρχικών αναγών της, ε, των αεροπορικών δυνάμεων του Αφγανιστάν. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα κάνουμε στα πλαίσια ενιαίας ε, αντιμετώπισης και χορήγησης εκπαίδευσης προς τις δυνάμεις του Αφγανιστάν. και το ΝΑΤΟ εδώ έχει εκφράσει την ευαρέσκειά του για τη συμμετοχή των δυνατοτήτων ε, της EDA. Σχετικά τώρα με την ε, κοινού χρήση, απόκτηση ε, των αεροπορικών μέσων. Αυτό θα βοηθήσει και την κάλυψη των μεμονωμένων αναγκών των κρατών μελών, θα καλύψει τις επιμέρους ανάγκες και εδώ στην τελευταία διαφάνεια μπορείτε να δείτε ποια θα είναι η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ποια η μεθοδολογία για την διασφάλιση της κοινή απόκτησης και ε, κοινή χρήση των μέσων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτερ Μπίλινγκ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αξιότιμους φουλευτές που μου έδωσαν την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιόν σας εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγομαι Πίτερ Μπίλινγκ και είμαι υπεύθυνο του τμήματος ε, για τις ε, επιχειρήσεις του λεγόμενου MIC, Monitoring Information. Θα μιλήσω σύντομα σήμερα για τις στατικές μεταφορές ως μέσον ε, χρήσιμο στην ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση καταστροφών. Θα, θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε τρία θέματα, βασικές αρχές για την χρήση των στρατιωτικών μέσων στην αντιμετώπιση καταστροφών. Δεύτερον, παράδειγμα σχετικά με το πώς εφαρμόσαμε πραγματικά την χρήση αυτής στρατιωτικών μέσων επιτόπου, δηλαδή για την αντιμετώπιση του πυλώνα στο Πακιστάν, σε αρχές του 2010. Και τρίτον, ορισμένες σκέψεις που κάνουμε για την βελτίωση πρόσβασης και χρήση των στατιωτικών μέσων και ικανοτήτων. Πρώτο λοιπόν τώρα μέρος της ε, παρουσίασή μου. Υπάρχουν εδώ ορισμένες ε, σημαντικές βασικές αρχές, καθώς και έγγραφα, όπω ε, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την ε, ε, βοήθεια. Έγγραφο του 2006, Military Support στην ε, αντιμετώπιση καταστροφών. Επίσης σημαντικό έγγραφο, το Oslo NTMC Guidelines, που επίσης έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτών των τριών εγγράφων, οι τρεις βασικές αρχές. Πρώτο, στρατιωτικά μέσα και ικανότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιορισμένες περιστάσεις και ως ίστατη καταφυγή. Αυτό σημαίνει όπου δεν υπάρχει συγκρίσιμη πολιτική ικανότητα για την αντιμετώπιση των ε, ανθρωπιστικών αναγκών. Δεύτερον, βασική ευθύνη των αρμόδιων αρχών είναι, είναι η ευθύνη των αρμόδιων αρχών της εθιγόμενης χώρας ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ε, συντονίζει ε, και αυτή η ευθύνη οφείλεται να γίνεται, οφείλει να γίνεται σεβαστή. Τρίτο, τρίτη βασική αρχή, η χρήση των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων πρέπει ωστόσο να σέβεται και να διατηρεί τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Αυτές λοιπόν είναι οι ε, συνθήκες πλαίσια υπό τα οποία λειτουργούμε στην αντιμετώπιση ε, καταστροφών και ανθρωπιστικών αναγκών. Δεύτερο μέρος της παρουσίασής μου, πώς τα εφαρμόσαμε τα πράγματα αυτά επιτόπου στο πεδίο. Πράγματι, οι στατιωτικέ ικανότητε μπορούν να είναι χρήσιμε για την αντιμετώπιση ε, καταστροφών ή ανθρωπιστικών αναγκών. Παράδειγμα, στην πράξη το Πακιστάν, ορισμένα πράγματα ήδη λέχθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, από ορισμένους από αυτούς, κατά βάση πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα των στρατηγικών αερομεταφορών. Αυτό έγινε με τριπλό τρόπο. Η ανθρωπιστικων αναγκων παραδειγμα στην πραξη το πακισταν ορισμενα πραγματα ηδη λεχθηκαν απο τους προηγούμενου ομιλητέ, απο ορισμενου απο αυτού, κατα βαση πώ αντιμετωπισαμε το θεμα των στρατηγικων αερομεταφορων αυτο εγινε με τριπλο τροπο η στρατηγικη μας πρώτα βασίστηκε στον εντοπισμό και ταυτοποίηση πολιτικών ικανοτήτων αερομεταφοράς που μπορούσαν να γίνουν είτε με pooling είτε με sharing ανάμεσα στις χώρες μέλη είτε μέσω της συγχρηματοδότησης με τα ε, μέσα που έχουμε για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών. Από το 2007 μέσα στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέχρι ενός ποσού 50% ε, τέτοιες επιχειρήσεις ε, μεταφορών. Βασικό όργανο μας αυτό, σε αυτό δόθηκε βέβαια η προτίμηση από την αρχή. Δεύτερη προτεραιότητα, εάν δεν μπορούμε ε, να εντοπίσουμε ή ταυτοποιήσουμε συγχρηματοδοτούμενες ή κοινή χρήση ικανότητες ή μέσα, στρεφόμαστε στους συναδέλφους μας του πυρήνα στρατηγικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στρατηγός τα είπε πριν αυτά, ζητήσαμε την υποστήριξή τους κατά τα μέσα Αυγούστου και μπόρεσαν πράγματι να εντοπίσουν τρεις δυνατότητες, τρεις ικανότητες μεταφοράς αν κόστους, δύο Αντόνοφ και ένα C17 ή ένα Αντόνοφ και δύο C17. για να το κάνουμε αυτό, για μας ήταν πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε τις στρατιωτικές αυτές ικανότητες, ωστόσο θα προτιμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, πολιτικού τύπου αεροσκάφη, έστω και αν είναι ναυλωμένα από στρατιωτικές αρχές. Και δύο από τα αεροσκάφη αυτά ήταν ε, πολιτικά. Τρίτο βήμα, εάν ούτε οι χρηματοδοτικές ικανότητες, ούτε οι ικανότητες για το MPC υπάρχουν, τότε στρεφόμαστε στους συναδέλφους μας του ΝΑΤΟ και δύο από τις 15 επιχειρήσεις συνολικά που συντονίσαμε προς το Πακιστάν έγιναν με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Μια μεταφορά πολλών τόνων ε, ε, μέσων υποστήριξης από την Σλοβακία και άλλες 40 παλέτες από τη Γερμανία στο Πακιστάν. Όλα αυτά γίνονται με πλήρη σεβασμό των κατευθυντήριων γραμμών του Όσλο έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο ο χώρος ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η ουδετερότητα της ανθρωπιστικής ε, δράσης, ιδίως σε δύσκολες περιστάσεις όπως αυτές ε, στο Πακιστάν. Αυτά είναι σκέψεις οι οποίες ε, πρέπει οπωσδήποτε να κυριαρχούν. Επίσης, ένα άλλο σχόλιο είναι σημαντικό. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι πάντοτε η έλλειψη διαθεσιμότητας ε, μεταφορικών ικανοτήτων έχουμε δει να υπάρχουν στην αγορά οι βασισμένες στην αγορά ικανότητες έχουμε για παράδειγμα ένα ε, μια σύμβαση μεσάζοντος που μας είχε εντοπίσει έξι τέτοιες δυνατότητες είναι θέμα όμως και χρηματοδοτήσεως οι χώρες μέλη βέβαια που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες που δεν έχουν τους απαραίτητους προϋπολογισμούς υφίσταται τον πειρασμό περισσότερο να χρησιμοποιήσουν τις δωρεάν προσφορές υποστήριξης από τους στρατιωτικούς αντί να χρειάζεται να καταβάλουν το 50% της συγχρηματοδότησης από την πλευρά τους. Αυτό λοιπόν επίσης πρέπει να εξεταστεί. Το τρίτο στοιχείο τώρα της παρουσίασής μου έχει ως εξή Πώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την χρήση των στρατηγικών ικανοτήτων αερομεταφορών. Εγώ συμφωνώ απολύτως με την ε, παρέμβαση του ταξιάρχου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΜΙΚ και MTC που ε, είναι επιτυχής και που συνεχίζεται. Μεταξύ άλλων έχουμε κάνει και εκπαιδεύσεις των αξιωματικών του MTC για την χρήση. Έχουμε προβλέψει επίσης και μια ε, συνάντηση για την άρση συμπερασμάτων, για την άρση διδαγμάτων από την εμπειρία μας μέχρι τώρα, ιδίω στο Πακιστάν. Ορισμένα από τα στοιχεία που ίσως προκύψουν ή μάλλον που ίσως τεθούν υπό συζήτηση είναι πρακτικά στοιχεία, δηλαδή ποιος αναλαμβάνει την φόρτωση και εκφόρτωση, ποιος ε, εξασφαλίζει την ε, real-time follow-up, την παρακολούθηση σε real-time των κινήσεων, πώς βελτιώνεται η ευκαμψία του συστήματος και εν τέλει πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο θέματα κόστους. Σε ορισμένα πλαίσια, για παράδειγμα, ίσως είναι χρήσιμο να εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφορά σε διαθαλάσσεις, όταν δηλαδή πρόκειται για ε, αγαθά μεγάλου όγκου που δεν είναι ίσως απαραίτητο να μετακινηθούν με τόση μεγάλη βιασύνη. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό follow-up, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στις 26 Οκτωβρίου, όπως λέχθηκε και πριν, όπου προτείνει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλουστευθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία για το pooling και co-financing και συγχρηματοδότηση δηλαδή των ε, ικανοτήτων και μέσων με χρήση των όσων προέρχονται από την ιδιωτική αγορά. Επίσης ο ιδιωτικός τομέας ε, να προσφέρει, να, να δηλώσει ποιες δυνατότητες υπάρχουν, να χρησιμοποιηθεί πλήρως το, η συμφωνία πλαίσιο για τις μεταφορικές ικανότητες καθώς και τα εργαλεία CSTP και τέλος, τέταρτο μάλλον, να συνεχιστεί η υποστήριξη για την ανάπτυξη ίδιας ικανότητας στρατηγικής αερομεταφοράς και για, για τη μετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών, καταστροφών κλπ. και μέσα στα πλαίσια των ΗΠΑ. Και αυτά βέβαια συζητούνται σήμερα και θα τελειώσω τονίζοντας δύο θέματα συντονισμός στρατιωτικού και πολιτικού τομέα που μπορεί να είναι κρίσιμος για την αντιμετώπιση καταστροφών. Χρειαζόμαστε τον συντονισμό, χρειαζόμαστε διευκόλυνση του συντονισμού με διάλογο, με ε, την σύνδεση, με προετοιμασία πριν να προκύψει η καταστροφή, η ηθομηνία. Δεύτερο βασικό συμπέρασμα, η Κομισιόν και ιδιαίτερα το ΕΚΟ, είμαστε ανοιχτοί στην χρήση στρατιωτικών μέσων για στρατηγικές αερομεταφορές αρκεί να τηρούνται αυστηρά οι κατευθείας γραμμές του Όσλο να μην συγχέονται τα όρια μεταξύ στρατιωτικού και, μη, και πολιτικού δηλαδή ε, τομέα και δράσης. Επίσης η ε, αποτελεσματικότητα πλευράς κόστους η κρίση για το αν είναι προτιμότερο να κινηθούν τα αγαθά είτε τα μέσα ε, εναερίως είτε θαλασσίως και επίσης η αντιμετώπιση επιτόπου των ε, καταστροφών ή θεομηνιών. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλινγκ, όλους ε, τους πυρογνωμονες και τώρα είναι η στιγμή για να τεθούν ερωτήματα. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους κύριοι μου για τις ε, πλήρεις <clears throat> παρουσιάσεις σας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε ίσως όλοι να τα επεξεργαστούμε και <clears throat> θα ήθελα να σας ζητήσω, εάν είναι δυνατόν, οι παρουσιάσεις σας με, το, με PowerPoint να δοθούν και στη γραμματεία για να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε πιο πολύ προσοχή στη συνέχεια. Θα ήθελα τώρα από πολιτική έποψη να πω ότι και η δική μου πολιτική ομάδα ότι θέλουμε να υπάρξει αυτή η συνεργασία, να υπάρξει συνεργασία μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα, αλλά επίσης και καλύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, καλύτερη από κοινού χρήση και διαμοιρασμός μέσων και ικανοτήτων από πραγματιστικούς ε, λόγους, αλλά και γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές από οικονομική άποψη και είναι απαραίτητο να υπάρξει σωστή χρήση των πόρων και καλή συνεργασία πολιτικού και στρατιωτική, πολιτικής και στρατιωτικής πτυχής, η οποία θα οδηγήσει και σε εξοικονόμηση αλλά και σε πιο αποτελεσματική χρήση των υπαρχουσών ικανοτήτων. Η νέα συνδίκη Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο μόνιμη μορφή συνεργασίας και επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε και περισσότερες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Έχω τώρα ορισμένα ερωτήματα, τώρα απευθύνονται σε όλους σας συλλήβδιν. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να αντιμετωπίσει το κάθε θέμα. Για τα θέματα των θαλασσίων μεταφορών εξεπλάγει λιγάκι ότι υπάρχουν καταρχήν κράτη τα οποία συμμετέχουν και τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά ακτογραμμές. Δεν είναι αρνητικό αυτό, απλώς με εκπλήσει το γεγονός ότι οι χώρες αυτές οι οποίες δεν είναι παράκτιες μπορούν να συμμετέχουν σε ενέργειες θαλασσίων μεταφορών. Επίσης για τον Ευρωπαϊκό Στόλο Εναερίων Μεταφορών, Αερομεταφορών και για την ε, δίκηση για τα θέματα αυτά. Εγώ εγώ βλέπω ότι υπάρχουν τέσσερις χώρες μέλη οι οποίες συμμετέχουν, ενώ είναι πολύ περισσότερες χώρες οι οποίες θέλουν στη συνέχεια να συμμετάσχουν στον ε, στόλο αυτό, στην συμμετοχή στο στόλο. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι χώρες αυτές δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο φορέα αυτό, αλλά θέλουν να συμμετάσχουν στο στόλο. Και ένα ακόμα ερώτημα για την ευρωπαϊκή διοίκηση ε, ε, Εναριο μεταφορών που βρίσκεται στο Eindhoven και επίσης <clears throat> και ο φορέας αυτός για την κίνηση και τις μεταφορές που βρίσκεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Βρίσκονται όλοι αυτοί σε ένα κοινό υπάρχει μια γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ των ατόμων αυτών, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους σε καθημερινό επίπεδο. Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Και για τις λεγόμενες diplomatic clearances, τις διπλωματικές διευκολύνσεις για τις στρατιωτικές αερομεταφορές. Εμείς έχουμε επιληφθεί του θέματος των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων και έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο ενιαίο για, τους, για τις πολιτικές αερομεταφορές, ώστε να μπορούν να κινούνται τα αεροπλάνα με ένα λογικό τρόπο και όχι ελίγδιν ή τη Ζίξαρτ. Ε, τι συμβαίνει όμως τώρα με τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Εσείς αναφερθήκατε σε ε, αποκλειστικές στρατιωτικές ζώνες που θέλετε να δημιουργήσετε για τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Τι θα συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουν πάλι παράκαμψη αυτών τα πολιτικά αεροσκάφη. <clears throat> Στην περίπτωση της ε, Γερμανίας έχει υπάρξει ουσιαστικά συγχώνευση του χώρου εποπτείας των πολιτικών αεροσκαφών και του χώρου των στρατιωτικών αεροσκαφών. Είναι η πρόθεσή σας να ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα και να μην είναι απόλυτα και χωρισμένοι αυτοί οι χώροι. Δηλαδή, εφόσον είμαστε όλοι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε όλοι τις καλύτερες δυνατές προθέσεις, μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο ενιαία εποπτεία <clears throat> και του πολιτικού και του στρατιωτικού χώρου και επομένως να μην χρειάζεται να έχουμε κλειστές περιοχές ε, για τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Δεν θέλω μόνο πολύ στο διάλογο, θα ήθελα να περιοριστώ λοιπόν σε αυτές τις παρατηρήσει. παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλωστε δεν έχουν μείνει και πολλοί βουλευτές πλέον. Ε, χαίρομαι που έχετε τον χρόνο να απαντήσετε σε ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να, να παρατηρήσω πρώτα ότι μου φαίνεται στενά χώρο μια τόσο σημαντική ε, συζήτηση να γίνεται με παρουσία τόσο λίγων ευρωβουλευτών. Ο κ. Γκάλερ είπε ήδη εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής του ομάδας ότι πολιτικά επιθυμούν να δουν την ε, στρατιωτική πολιτική συνεργασία, την θεωρούν πολύ θετική. Η δική μου ε, πολιτική ομάδα, η Ενωτική Αριστερά, σε πολλά σημεία στέκεται πολύ κριτικά απέναντι στην συνεργασία αυτή. Ήδη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ορισμένοι από τους άλλους ομιλητές είπαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές ικανότητες μόνον εφόσον δεν υφίστανται οι πολιτικές. Κατέστη σαφές ποιες είναι οι στρατιωτικές ικανότητες που υπάρχουν, ποια εφέ, ποια ε, αποτελέσματα συνέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες αυτές τις λέξεις, sharing, pooling κτλ. Δεν θα τα επαναλάβω εγώ και κατέστηκε σαφές και ποιο είναι, ποια είναι η πίεση κόστους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα ποιος βοηθάει στο μέλλον ποιον. Αφενός είναι σαφές ότι μέσα στα πλαίσια του θετικού τομέα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποιες ε, συνέργειες, κάποια synergy effects δηλαδή, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και η στρατιωτικοπολιτική συνεργασία θα προσφέρει και κάποια νομιμοποίηση ώστε να περάσουν περισσότερα χρήματα και στο στρατιωτικό τομέα. Να καταλήξουν δηλαδή περισσότερα κονδύλια στο στρατιωτικό τομέα. Δεν είναι σαφές για μένα λοιπόν γιατί δίνονται περισσότερες ικανότητες στο εκδικό τομέα, προσφέρονται εν τέλει, και λιγότερο στον ανθρωπιστικό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρόκειται να αυξηθούν αυτές οι ικανότητες με τον τρόπο που εξήγησα. Από εκεί ξεπηδά και το ερώτημά μου, εάν υπάρχει κάποιο κενό κάλυψης σε ό,τι αφορά καθαρά τις πολιτικές ικανότητες μεταφορές, αν υπάρχει δηλαδή κάποια έλλειψη, κάποιο έλλειμμα και πόσο μεγάλο είναι αυτό. Πριν να προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτών των ε, συνεργειών, προτιμώ να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να ρωτήσω επίσης, τι θα γίνει εάν για παράδειγμα, τύχη στρατιωτικά, στρατιωτικά αεροσκάφη να απαιτούνται ταυτόχρονα για την υποστήριξη μιας στρατιωτική παρέμβασης αλλά και για την αντιμετώπιση, αλλά σε άλλη χώρα, μιας ανθρωπιστικής επίγουσα κατάστασης. Πού θα δοθεί η προτεραιότητα όταν υπάρχουν τόσο πολλές ικανότητες ε, στο στρατιωτικό τομέα. Και η τελευταία μου ερώτηση αναφέρεται στις κατευθυντήρες γραμμές του Όσλο που τις ανέφερε κατ' επανάληψη ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν. Γενικά επιδιώκεται αυτή η ε, στενότερη συνεργασία. Η χρησιμοποίηση τακτικών αεροσκαφών σίγουρα θα αποτελούσε ένα βήμα για περαιτέρω τέτοια συνεργασία η δημοσίευση της Κομισιόν που λέει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ικανότητας αντιμετώπισης ανθρωπιστικών καταστροφών και το 2010, έτσι λέει το έγγραφο αυτό, ε, τονίζει ε, περισσότερο την ανάγκη συνεργασίας για αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ε, αναγκών με ενδεχόμενες επιχειρήσεις που δρούν ήδη επιτόπου. Αλλά συχνά αυτές δεν είναι, αυτές οι επιχειρήσεις δηλαδή, δεν είναι ουδέτερες, αλλά έχουν συμπαραταχθεί με τη μια ή την άλλη πλευρά ενός εμφύλιου πολέμου. Αυτό στην πραγματικότητα παραβιάζει, κατά τη γνώμη μου, τις ε, γραμμές του Όσλο, που απαιτούν απόλυτη ουδετερότητα, αυστηρή ουδετερότητα, και που είχαν γίνει δεχτές ως βάση από το 2007 για τις ενέργειες αυτές. Τώρα, ερώτηση προς την Κομισιόν, αλλά και προς τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου εδώ πώς αντιμετωπίζουν τον προβληματισμό αυτό. Thank you Σας ευχαριστώ. Ας απαντήσετε με την σειρά που κάνατε τις ε, ε, παρεμβάσεις σας. Μπορείτε να απαντήσετε σε όποιε ερωτήσει θέλετε, αλλά παρακαλώ μην απαντήσετε, μην μακρηγορήσετε, όχι περισσότερο από πέντε λεπτά. Κύριε Παυλόπουλο, εσεί. Αν με συγχωρείτε, υπάρχει ακόμη μια ερώτηση από τον κύριο Στάσνη. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ενημερωτική και χρήσιμη η συζήτηση αυτή για την κατεύθυνση όπου κατευθυνόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Ένωσης με χρήση των υφισταμένων ικανοτήτων και ελπίζω όλοι, όλες οι πλευρές να ωφεληθούν. Οι ανησυχίες μου είναι παρόμοιες με αυτές του συναδέλφου μου Μίχαελ Γκάλερ. Είδα την European Transport Command Ξέρω ότι είναι πολύ νέος ο οργανισμός αυτός και ελπίζω να αναπτυχθεί. Όπως ο κύριος Γκάλερ και εγώ δύσκολα βλέπω πώς είναι δυνατόν εσωτερικές έγκλειστες χώρες να συμμετέχουν στις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά η Σλοβακία, για παράδειγμα, μπορεί να συμμετάσχει στο European Air Transport Center και να υπάρξει και συμμετοχή και εμπλοκή και άλλων χωρών. Για την ώρα φαίνεται η προσπάθεια αυτή να ε, εστιάζεται περισσότερο στο κέντρο και στο βορρά, με χώρες Μπενελούξ, Γερμανία κλπ. Αλλά υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν και άλλες πλευρές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν και αποτελεσματικότητα και ικανότητες. Και επίσης η ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τη χρήση του ενέργειου χώρου. Ελπίζω με το νέο σύστημα πλοήγησης ΣΥΖΑ να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικούς καιρούς και όλοι αυτοί οι κατασκοπικοί δορυφόροι ε, τέλος πάντων τα αεροσκάφη και τα πολιτικά αεροσκάφη που περνούν πάνω από ε, εναέριους ε, ε, στρατιωτικούς εναέριους χώρους εκεί δηλαδή όπου είναι βάση κλπ δεν πρόκειται να προκαλέσουν ζημιά ελπίζω ότι το σύστημα αυτό θα προσφέρει τις λύσεις και ίσως μπορείτε να σχολιάσετε τα θέματα αυτά Thank you Ευχαριστώ. Εσείς, Δίαρχη. Sir, uh, Mr. if I have... Uh, Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Το βασικό πράγμα το οποίο προσφέρει το Κέντρο Συντονισμού ε, Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών προς τα μέλη του είναι ότι ακόμα και για χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν ε, σύνορα με τη θάλασσα και δεν έχουν ε, θαλάσσια μέσα, τους προσφέρουμε ακριβώς τα θαλάσσια αυτά μέσα. Οι Έλληνες εφοπλιστές με τους οποίους συνεργαζόμεθα έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη στιγμή το 18% του παγκόσμιου στόλου εμπορικών μεταφορών. Oh, Σχετικά με το ATC και το CEE κάθε φορά τίθονται, τίθενται συγγνώμη, ερωτηματικά γύρω από το στόχο που έχουμε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβετε είναι ότι το ATC είναι ε, κάτι που ασχολείται με τα στρατιωτικά μέσα για τις αερομεταφορές. Το ATF είναι ένα δίκτυο κρατών, στρατιωτικό αρχηγείο τι σημαίνει. Και γι' αυτό είναι μοναδική η περίπτωση αυτή, ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση για τη δημιουργία του στρατηγίου αυτού, περιμένουμε ακόμα και το Βέλγιο βέβαια, είναι κάτι που δεν συμβαίνει στα πλαίσια του MCC ή του ATF, που είναι απλά θέματα συντονισμού. Σαν παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο αυτό έγινε μια επιχείρηση η οποία ήταν απόλυτα ελεγχόμενη Ε, ενέργεια από εμά που είχε να κάνει από το Eindhoven που είχε να κάνει με μεταφορά ατόμων από το κέρας της Αφρικής στην ε, Ολλανδία. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία πτήση <clears throat> στην Αφρική με γερμανικά ε, πληρώματα. Εμείς ουσιαστικά είμαστε μια υπηρεσία που ελέγχει τις αποστολές. Γι' αυτό λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο και δεν χρειάζεται να επαρχόμεθα στα κράτη-μέλη για να ζητούμε ε, συγκεκριμένες ε, ενέργειες. Το ATIS είναι μια στρατιωτική βέβαια δομή και το MCCE έχει μια σαφή αποστολή. Όλο και περισσότερο εμείς έχουμε ένα φόρτο εργασίας ο οποίος έχει να κάνει με τη συνεργασία των τεσσάρων κρατών <clears throat> μεταξύ των τεσσάρων χωρών τα περισσότερα από τα αεροσκάφη ήδη έχουμε την ε, έγκριση να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα θέσουμε σε αποστολές. Αλλά το MCC, όπως ξέρετε, εμπλέκει και περισσότερες χώρες. Και πάλι σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν η Γαλλία ζητά από το ATC να προχωρήσει σε μία αερομεταφορά, εμείς κοιτάμε <coughs> ποιες είναι, ποιοι είναι οι σχηματισμοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και αν δεν είναι επαρκούν χρησιμοποιούμε το MCC για να μπορέσουμε να βρούμε περαιτέρω μέσα. Είναι διαφορετική λοιπόν η, λειτουργία του ATC με το MCC. Αλλά συνεργαζόμαστε. Υπήρξε και ένα, ερώτημα για τη διεύνηση σε περαιτέρω κράτη-μέλη για το MCC. Εμείς χρειαστήκαμε πάνω από 11 χρόνια για να εδραιώσουμε το MCCE και το πρώτο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε είναι να έχουμε μια ανθεκτική δομή διοίκησης προτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω ε, διευρύνσεις. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αναρμονίσουμε τις διαδικασίες να υπάρχει μια πραγματική ενιαία διοίκηση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικέ διοικήσει, Αλλά η βασική αυτή δομή των τεσσάρων που εμπλέκει τέσσερα, χρό... τέσσερα κράτη θα πρέπει να δει πώς θα μπορέσει να τα φέρει σε πέρα όλα αυτά για περισσότερα κράτη. Ε, Mr. Ε, Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Καντέν. Ευχαριστώ, θέλω να θίξω το θέμα του γιατί μια χώρα που δεν έχει ε, ακτογραμμή χρειάζεται θαλάσσιες μεταφορές και επίσης να συνεχίσω αυτό το οποίο ελέγχθη, την διαδραστική επιφάνεια μεταξύ MCC και EATF. Στο ΝΑΤΟ έχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο φιλοδοξίας. <clears throat> Ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές στον κόσμο όπου πρέπει να αναπτύξουμε δυνάμεις και ικανότητες. Και ποιες είναι οι ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν φυσικά για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στις διαδικασίες σχεδιασμού μας βλέπουμε τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και λέμε ποιες είναι οι ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και επομένως επιμερίζουμε αυτό στα διάφορα κράτη-μέλη. Και εδώ επιμερίζεται και η ικανότητα θαλασσίων μεταφορών και αερίων μεταφορών και γι' αυτό χώρες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα είναι υποχρεωμένες και αυτές να συμβάλλουν στις θαλασσίες μεταφορές. Παραδείγματος χάρη η τσεχική δημοκρατία έχει μετακινήσει μέσα στο Αφγανιστάν με συνδυασμένη ε, μεταφορά διαξηράς και μετά δια Είναι πιο απλό να μεταφέρει κανείς πράγματα και εξοπλισμό δια θαλάσσης παρότι με αερομεταφορά. Επομένως βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ταυτοποιήσουν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και το κατά πόσο είναι πρόσφορο να γίνει θαλάσσια μεταφορά. Αλλά για τα κράτη τα οποία έχουν <clears throat> συμμετοχή στις ομάδες μας, συζητούμε από τις, ομάδες, από τις χώρες αυτές ή να αποκτήσουν μέσα θαλασσίων μεταφορών ή να συμμετέχουν στο MCC e και επομένως να αρρωγήσουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία μεταφέρουν ε, μέσα και εξοπλισμό είτε εναερίω είτε διαθαλάσσια. Ακόμα λοιπόν και μια χώρα που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα πρέπει να έχει την ικανότητα θαλασσίων μεταφορών. Για την σχέση του ATC και του MCCE, αν δείτε το ιστορικό, όπως το ανέφερα ε, στην ε, παρουσίασή μου, υπήρξαν κάποια προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν Ήδη από το 1989 υπήρξε μια ειδίκευση ομάδων σε κρατών άλλων σε αενάριες μεταφορές και άλλες σε θαλάσσιες μεταφορές. Και μετά είπαμε γιατί να μην συνδυάσουμε τις δύο αυτές ε, δομές και να μπορούμε να λειτουργούμε από κοινού. Και αυτό έγινε και γι' αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τα δύο κέντρα είναι πλέον συν, συγχωνευμένα μεταξύ τους και σιγά σιγά και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ορισμένα κράτη συγγνώμη, από το ΝΑΤΟ έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στι ικανότητέ του και γι' αυτό έχουν δημιουργήσει το ATC. Το MCC είναι αυτή τη στιγμή μια ομάδα βασικά τεσσάρων κρατών που έχουν πολύ λιγότερα προβλήματα εσωτερικού συντονισμού και μπορούν να συνεργάζονται με τα άλλα κράτη. Αυτό το οποίο είναι κεφαλαιόδες είναι να υπάρξει ο διαμοιρασμός πληροφοριών, αλλά φυσικά και ανθρώπινου υλικού, γιατί δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι ειδικοί για τα θέματα μεταφορών και μετακίνησης ε, υλικού και δεν θέλουμε να τους χάσουμε και να φύγουν από το MCC και να πάνε στο ATC στο μέλλον, αν οι δύο φορείς αποφασίσουν να κινηθούν τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Είμαστε λοιπόν απόλυτα ανοιχτοί στο να είμαστε στον ίδιο χώρο ή να έχουμε άλλες μορφές συνεργασίας για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό που είναι απαραίτητο να υπάρχει αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο στρατηγός Πούρη. Πάρα πολλά θέματα, απλώς θέλω να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα <clears throat> ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ κρίσιμο θέμα η συνεργασία Πολιτική πτυχή και στρατιωτική πτυχή και εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την συνέργεια μεταξύ τη στρατιωτική και μη στρατιωτική ικανότητα. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ήδη από την 1η Ιανουαρίου όταν η υπηρεσία εξωτερικής δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πλήρω ενεργή, ότι θα προέλθει και κάποια επιτάχυνση στη διαδικασία αυτή. Θέλω να τονίσω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο ίσω δεν υπογραμμίστηκε αρκετά, είναι το θέμα τη εκπαίδευση η εκπαίδευση την οποία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μαζί με το ΜΙΚ βαίνει όλο ένα βελτιούμενη. Μεταξύ της 14ης και 18ης Μαρτίου του 2011 θα λάβει η χώρα μια άσκηση για ανακουβιστικές ενέργειες η οποία θα γίνει στο Μανάτο στην Ινδονησία και θα συμμετέχει η UNPC, το, η Movement και η Transportation θα συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση. Αυτή λοιπόν είναι μια άσκηση η οποία θα εξασφαλίσει ακόμα καλύτερη συνεργασία με την ΜΙΚ στα θέματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μουτσιάκης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο συσχετισμός του ATF και του ATC των δράσεών τους και των στόχων τους είναι κάτι το οποίο έχει ήδη απαντηθεί από τον κύριο Ρουσό. Το ATC, όπως υπόθηκε, είναι στην ουσία ένα λειτουργικό αρχηγείο, επιχειρησιακό αρχηγείο, ενώ το ATF είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε 15 χώρες μέλη που έχουν υπογράψει την επιστολή προθέσεων. Σας είπα επίση ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν επικαλύψεις. Σαν παράδειγμα, το επόμενο πρόγραμμα συνάντησης θα οργανωθεί στο ATC, στους χώρους του ATC και θα υπάρχουν ε, διασταυρούμενες κοινέ ενημερώσεις, briefings για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή επικάλυψης. Το ATC θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στα πλαίσια του ATF για να αποφύγουμε όπως είπα τις επικαλύψεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχάς το επιχειρησιακό στρατηγείο το οποίο είναι ήδη ισχυρό και από την άλλη έχουμε το πλαίσιο συνεργασίας. Επιπλέον να πω ότι αρχικά Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό σχετικά με τον καθορισμό των στόλων, πιστεύαμε ότι το ATC θα ήταν το επιχειρησιακό στρατηγείο του ATF. Αλλά τώρα είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας και δεν υπάρχει μια τέτοια σχέση πλέον. Το δεύτερο θέμα σχετικά με τις διπλωματικές διευκολύνσεις για τις ε, στρατιωτικές πτήσεις και αν θα βασίζονται και θα περιορίζονται στις στρατιωτικές περιοχές που έχουν ε, κλείσει. Αυτό θα γίνεται στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού σε εισαγωγικά. Σχετικά τώρα με τη στρατιωτικά αεροσκάφη και με ποιο τρόπο ε, θα επηρεαστούν από το σύστημα αυτό του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού οι στρατιωτικές πτήσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας και θα κατατεθούν τα πρώτα συμπεράσματα στην επόμενη συνάντηση. Έχουμε επίσης υποβάλει και συστάσεις και στα πλαίσια της ε, Διοικητικής Επιτροπής του ΝΑΤΣ, σχετικά με τους, ε, όπου συμμετέχουν οι γενικοί διευθυντές. Η διαχείριση των αεροπορικών μεταφορών δεν καλύπτεται από την υπηρεσία. Εμείς ασχολούμεθα μόνο με τις ε, διπλωματικές διευκολύνσεις, τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπίλινγκ τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε υπήρξε μία ερώτηση σχετική με τις κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο και πώς θα αντιμετωπιστούν εφόσον υπάρξει μία αποστολή e SDP και μία ανθρωπιστική επίσης αποστολή ταυτόχρονα. Οι κατευθυντήριες ε, του Όσλο είναι ιδιαίτερα σοφές εδώ, βασίζονται στην εμπειρία και μερικές φορές εμπειρία ιδιαίτερα δυσάρεστη. Λοιπόν, εφόσον εμείνουμε στο σεβασμό των αρχών αυτών, τα πράγματα θα πάνε καλά. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς οι επιχειρήσεις θα αναλαμβάνονται στο μέλλον. Σαν παράδειγμα, κρίση είναι μια φυσική καταστροφή, είναι κάτι το πιο περίπλοκο Νομίζω ότι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τη στρατιωτικά μέσα με τον ένα τρόπο ή τον άλλο είναι κάτι το οποίο είναι προσυζήτηση. Ή είναι απλά ένα θέμα καταστροφής στην Ευρώπη. Από την άλλη ένα άλλο θέμα που είπατε είναι το κενό που υπάρχει, κενό επιχειρησιακό, κενό οικονομικό κενό σε επίπεδο χρονισμού, σε επίπεδο κατεπήγοντος. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να κριθεί το είδος της καταστροφής και το είδος της απάντησης που θα είναι διαθέσιμο. Πρέπει να αναπτυχθούν ξεκάθαρα κριτήρια και στο τέλος θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα κριτήρια αυτά κατά περίπτωση, να τα κρίνουμε μάλλον κατά περίπτωση προς όφελος νομίζω ε, κυρίως ε, των πιο ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, πώς μπορούμε εμείς να ωφελήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπου ανθρωπιστική βοήθεια να ωφελεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, αλλά παρόλα αυτά να υπονομευθεί αυτό από μια παρέμβαση στρατιωτικού τύπου που μεταφέρει κάποιες εκατοντάδες τρόφιμα και αυτό οδηγεί σε αναζωπήρωση σαν παράδειγμα ε, των συγκρούσεων ανάμεσα σε στρατιωτικές μονάδες επιτόπου. Νομίζω λοιπόν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν ξεκάθαρα κριτήρια. Υπάρχουν πάντα φαιές περιοχές βέβαια, είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσει κανείς ε, να αξιολογήσει σωστά ε, το τι ε, είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει για αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά όπως είπα στην αρχή, οι κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο μας παρέχουν τις βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την ε, ανάπτυξη των δομών σας και ελπίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον την ευκαιρία στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση και θα θέλαμε να έχετε ως τον πιο αποτελεσματικές δομές και όχι σε επίπεδο ανταγωνισμού ή επικάλυψης των υπηρεσιών αυτών. Έχουμε το επόμενο σημείο που αφορά τώρα την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε εδώ. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να ανταλλάξουμε απόψει για την... Έπρεπε να ανταλλάξουμε απόψει με τον κύριο Σάριου Βόλσκι, τον επικεφαλή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Δυστυχώ δεν, είναι, δεν μπόρεσε να είναι παρόν ο κύριο. Ε, ε, Σαρσβόλσκι. Έχουμε όμως την γραπτή έκθεση και έχουμε και τον κύριο Πάσκο, ο οποίος είναι ο, προ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια σε σχέση με αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Με παρουσιάζετε σαν να είμαι ο τελευταίος επιβι... επιβιώσας κάποιας ε, επιτροπής ή κάποιας ομάδας εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές ε, συνδιασκέψεις αυτού του είδους και ήμουν φυσικά και ο επικεφαλής της ρουμανικής αντιπροσωπείας. Μπορώ να σας πω ότι η εντύπωσή μου είναι ότι σε σχέση με προηγούμενες φορές αυτή τη φορά οι συζητήσεις ήταν πολύ πιο εστιασμένες, πολύ πιο επαγγελματικό το κλίμα και οι εκθέσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν επίσης στην ε, Επιτροπή Άμυνας που είναι αυτή στην οποία εγώ ήμουν παρόν, γιατί αυτή ήταν η αποστολή μου, ήταν καλές εκθέσεις και είχαμε θετικές συζητήσεις. Η θέση τώρα της Πολωνίας παρουσιάστηκε με αρκετά ενδελεχή τρόπο σε άλλες επιτροπές και ήταν μια πολύ καλά αρθρωμένη, διαθρωμένη θέση. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις ίσως ε, χρειάζεται περισσότερη εξέταση, περισσότερο, περισσότερη υποστήριξη. χάρη η πρόταση να υπάρχει μια Επιτροπή Ασφάλειας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τολμηρή πρωτοβουλία. Έτσι θεωρούσα, αλλά είδα μετά να κυκλοφορεί ένα έγγραφο που έλεγε ότι εγώ ήμουνα εναντίον του. Και επίση ο Σάρο Βόλσκι, ο οποίο δεν ήταν παρόν και αυτό φέρεται να ήταν εναντίον αυτή τη πρωτοβουλία. Δεν είπε απολύτω τίποτα. Ο κύριο Σάρο Βόλσκι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό το οποίο αναφέρεται σε κάποια έγγραφα. Αυτό παρενθετικά. Η Σύνοδος Ολομέλης επίσης αντιμετώπισε κάποια από αυτά τα ζητήματα υπήρξε μεγάλη συζήτηση με τον Αμερικανό πρεσβευτή με τη Μάτσια Ρίζ, συγγνώμη, την Αμερικανίδα πρεσβευτή η οποία ήταν αναπληρώτρια, αναπληρώτρια πρεσβευτής τουλάχιστον και έτυχε χρειάστηκε να απαντήσει πολλά ερωτήματα σε σχέση με την πολιτική της ε, Αμερικανικής κυβέρνησης. Κάτι το οποίο δεν έτυχε θετικής αποδοχής είναι ότι όπως ξέρετε ο κ. Ράσμουσεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μας μίλησε μέσω βιδεοδιασκέψεως. Δεν υπήρχε δυνατότητα διάδρασης. <clears throat> Αυτό ήταν μια ατυχή συγκυρία, μια κοινοβουλευτική συνέλευση η οποία λάμβανε χώρα συγχρόνως με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν μπορούσε να παρίσταται ο κύριος Ράσμουσεν, δεν μπορούσαμε να διακτηνήσουμε τμήμα του κύριου Ράσμουσεν ώστε να είναι μαζί μας στη Βασοβία, αλλά αν είχε υπάρξει μεγαλύτερη επιμονή θα μπορούσε να είχε υπάρξει μια διασύνδεση βίντεο που να επέτρεπε και τη διάδραση μεταξύ μας. Ο νέος πρόεδρος της ε, συνέλευσης της, ε, του ΝΑΤΟ, κ. Λάμερς, είπε ότι την επόμενη φορά θα είναι παρόν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με σάρκα και οστά. Επομένως την επόμενη φορά δεν θα έχει τρόπο να ξεφύγει από τη συνάντησή μας. Εν κατακλείδη νομίζω ότι ήταν μια επιτυχής συνάντηση. Όπως σας είπα δεν ήταν ευτυχής η συγκυρία <clears throat> της ε, χρονικής σύμπτωσης αυτής της συνάντησης με τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά ήταν ένα είδος προθέρμανσης εν μέρη και για τη διάσκεψη κορυφής για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη συνέχεια στη διάσκεψη κορυφής. Ε, ουσιαστικά μπορέσαμε να πιάσουμε το σφιγμό της διάσκεψης κορυφής και η τελική μου παρατήρηση είναι ότι για μια ακόμα φορά πρέπει να τονίσω ότι ήταν πολύ καλή η διοργάνωση και οι πολωνικές απόψεις παρουσιάστηκαν πολύ καλά και παρουσιάστηκαν από άτομα υψηλού επίπεδου. Και είχαμε έτσι την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις του Εθνικού ε, Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στην ε, Πολωνία και πιστεύω και σε άλλες επιτροπές που ήταν παρουσίαση τη συνδιάσκεψη υπήρξαν άλλοι υψηλοί εκπρόσωποι. Ήταν μια επιτυχή συνεδρία λοιπόν. Mr. Pascu, I would like to ask uh, the last... Uh, Θα ζητήσω τώρα στα υπολοιπόμενα μέλη της, Επι... Επιτροπής μας αν έχουν να θέσουν κάποια ερώτηματα. Ο Μάικελ. Όχι λέει ο Μάικελ. <clears throat> Αλλά μια πρόταση την επόμενη φορά. Γιατί να μην γίνεται μια μέρα πριν από τη διάσκεψη κορυφής που έγινε στη Λισαβόνα. Εμείς είχαμε πριν από τη συνεδρίαση στην Τριπολίτιδα μια συνάντηση με τον κύριο Πίμπαλξ που ήρθε στην Επιτροπή μας. Αν είχε γίνει κάπου αλλού η συνάντηση αυτή δεν θα μπορούσε να είναι παρόν. Λοιπόν, όταν γίνεται μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι παρούσα και η διακοινοβουλευτική συνέλευση και να έχει τη δυνατότητα να συνεδριάσει, να μην παραγνωρίζεται λοιπόν και γι' αυτό να κάνει μια συνάντηση μια μέρα ή δύο πριν από την ε, διάσκεψη εκτελεστικού χαρακτήρα του, ΝΑΤΟ. Ναι, και στη Λισαβόνα θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Λυπάμαι για την ε, ποιότητα του καιρού στην Πολωνία, λέει ο Προεδρεύων. Κύριε Στράσεν, θέλετε να πείτε τίποτα. Ε, εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είναι η τελευταία συνεδρίαση της υποεπιτροπή μας για φέτος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, τα μέλη, την γραμματεία, τους συνεργάτες, βοηθούς, διερμηνείς